Παρακαλώ καθίστε. Καλημέρα, είμαι η Πρόεδρος. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να αρχίσουμε με τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις. Πρώτο σημείο της ημερησίας διάταξης. Έγκριση της ημερησίας διάταξης. Δεν έχω προτάσεις τροποποιήσεις. Θα ήθελα να πω στους συντονιστές πως αναβάλουμε την αυριανή συνάντηση των συντονιστών στις 11. Αύριο θα τελειώσουμε στις 11. Δεν είμαι ικανοποιημένη με αυτό, αλλά κάποιοι συντονιστές δεν ήταν διαθέσιμοι. Μου το είπαν μόλις χθες το βράδυ. Γι' αυτό και λυπούμε πολύ γι' αυτό. Δεν έχω τις ημερήσεις διατάξεις. Θα ήθελα να υποδείξω πως το σημείο 45, 46 52 θα γίνει αντικείμενο ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα αντί για αύριο. Για το EDF σήμερα αντί για αύριο. Είμαστε αύριο αντί για σήμερα, συγγνώμη. Για το σημείο 2 της ημερησίας διαταξής θα ήθελα να πω πως οι γλώσσες, διαθέσιμες είναι οι γλώσσες που βλέπετε από το φυλάδιο όπως πάντα έχουμε μετάδοση της συνεδρίασης από το διαδίκτυο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να έχετε τις κάρτες ψηφοφορίας μαζί και στις 10 θα έχουμε ενός λεπτού σιωπή για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Βρυξέλλες πριν από ένα χρόνο εδώ, πολύ κοντά στο σημείο αυτό και στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Φτάνουμε στο σημείο 3, την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του ΕΤΣΕ, θα ασχοληθούμε με ένα σχέδιο γνωμοδότηση. Συζητητή είναι ο συνάδελφο Τάκουλα, ο οποίο σε λίγο θα πάρει τον λόγο. Για την παρουσίαση τη έκθεση θα ήθελα να καλωσορίσω τα δύο μέλη του Ελεκτικού συνεδρίου υπεύθυνα για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο. Καλώ ήρθατε, κύριε Τάκουλα. Αγαπητοί συνάδελφοι, Με μεγάλη μου χαρά τώρα λαμβάνω τον ε, ε, λόγο και θα σας μιλήσω στην πιο γοητευτική γλώσσα του κόσμου. Α, υπάρχει ένα πρόβλημα τεχνικό με την ε, μετάφραση. Ακούγεστε, μεταφράζεται. Δεν περνάει η αγγλική μετάφραση, λέει. Ε, Okei. näytetään, eikö ole, on, on tulkkaus vai eh. Λύθηκε το τεχνικό πρόβλημα. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσετε χωρίς πρόβλημα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Στάκουλα. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Πρόκειται για την ανάγκη της Ευρώπης να έχει κάποιες επενδύσεις. Είναι μια ιδέα που ξεκίνησε τη διαδρομή της το 2008 και από το 2008 έχουμε αυτό το λεγόμενο Ταμείο Γιούνκερ τα τελευταία δύο χρόνια. Την σήμερα ημέρα θα πρέπει να διαπιστωθεί ε, ε κατά πόσο θα έχουμε χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα ούτω ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για τις στρατηγικές επενδύσεις. Θα πρέπει επομένως να δούμε πώς θα γίνει και το εύση θα ε, γίνεται όλο ένα πιο αποτελεσματικό αλλά και θα διέπεται από μεγαλύτερη διαφάνεια. Θέλω επομένως στην ε, πρότασή μου να σταθώ σε τέσσερα στοιχεία. Πρώτα-πρώτα, τα σχέδια και προγράμματα του ΕΦΣΙ θα πρέπει να διακρίνονται από διαφάνεια όσο γίνεται περισσότερο. Επίσης, τα σχετικά κριτήρια για αυτά θα πρέπει να διέπονται από δημοσιότητα Οπότε έτσι πρόκειται να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των αγορών για τα σχέδια και προγράμματα του ΕΦΣΙ. Πρέπει να χαρακτηρίζονται αυτά από καινοτομία και έτσι να αποτελούν ε, μια ε, προστιθέμενη αξία. Οπότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το στοιχείο του κινδύνου. Να, δηλαδή αυτά που έχουν κάποιο στοιχείο κινδύνου Αυτά θέλουμε να χρηματοδοτηθούν ε, με αυτόν τον τρόπο γιατί αλλιώς δεν θα ετύχαναν χρηματοδότηση. Και έχουμε συνοηθεί με τον ε, Επίτροπο Κατάινεν για τις δυνατότητες που υπάρχουν της αξιοποίησης αυτών ε, των προγραμμάτων και είναι πάρα πολύ μεγάλες αυτές οι δυνατότητες. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα η σωστή κατανομή μεταξύ των χωρών. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε πως θα αξιοποιηθεί παντού η δυνατότητα που μας έχει δημιουργηθεί παντού, παντού στην Ευρώπη και στις πιο μακρισμένες περιοχές και επίσης στις πιο αραιοκατοικημένες. Οπότε έχουμε τώρα αυτά τα σχέδια, αυτά τα προγράμματα που θα πρέπει να διακρίνονται από σαφήνεια, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την αχρίαστη γραφειοκρατία. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που φύγω στο κείμενό μου και θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να δούμε την διαδικασία μετά από τον διάλογο και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να προσέξουμε αυτή την υπόθεση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σάρο μας ζήτησε το λόγο. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω, ίσως να μιλήσω φιλανδικά σήμερα. Αλλά δεν ξέρω, μην νομίζετε ότι είναι κάποια συνωμοσία. Τέλος πάντων. Πρώτα απ' όλα, να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή ε, για τα ξεκάθαρα μηνύματά του και σαφές ε, το τι θέλει. Να περάσουμε στα κύρια σημεία. Όλοι ξέρουμε το έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι πρέπει να είναι διαφανές ε, και ειδικά στην επιλογή των έργων. Επίσης, για την απλοποίηση της ε, διαδικασίας και για το ότι δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά έχω κάποιες επιφυλάξεις για την ε, γεωγραφική ανισορροπία που ανέφερε ο εισηγητής. Καλό είναι να το κοιτάμε αυτό, αρκεί να μην γίνει η ίδια η ανισορροπία το βασικό θέμα. Αν μπορούμε να δούμε το θέμα της ανισορροπίας και να υπάρχει μια καλύτερη γεωγραφική ισορροπία, όσο γίνεται βεβαίως κάτι τέτοιο χωρίς να αντιβαίνει στην αναγκαιότητα και στην κερδοφορία των επενδύσεων, τότε καλώς. Θα ήθελα τώρα εγώ να προσθέσω και να τονίσω και να υπογραμμίσω το ότι είναι λύπηρο το, ελεγκτικό, το ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει έναν αρκετά ισχυρό ρόλο, τον ρόλο που θα ήθελε δηλαδή. Στα χαρτιά τον έχουν και την πρώτη φορά φροντίσαμε το ελεγκτικό συνέδριο να έχει την πρόσβαση που ζητάει αλλά φαίνεται τα τελευταία χρόνια ότι στην πράξη υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να δούμε γιατί προφανώς το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι ικανοποιημένο 100% με την πρόσβαση που έχει. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά. Αυτά ήθελα να πω αυτή τη στιγμή. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσω να ρωτήσω τον εισηγητή, το ελεγκτικό συνέδριο. Α, α, συγγνώμη. Α, δεν σας είδα. Δεν σας είδα, κύριε Πυρίνσκι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Θεωρώ ότι αξιολογώντας την εφαρμογή του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου βεβαίως ε, την προσθετικότητα. Αυτό είναι ο λόγος ε, ύπαρξής του για να δούμε ακριβώς και σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται στις ε, προσδοκίες. Και εδώ πέρα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια πράγματα που είπε ο εισηγητής, δηλαδή την έκκληση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να σκεφτεί προσεκτικά την πραγματική προσθετικότητα και δυναμική. Αυτό είναι στην παράγραφο 13. Επίσης, ζητά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δώσει πληροφορίες για το φαινόμενο μόχλευσης ε, και όχι μόνο τον μέσο όρο που θα δείχνει το μέγεθος των ιδιωτικών κεφαλαίων που προσέλκυσε Επίσης η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων θα πρέπει να αξιολογείται με μια ποσοτικοποιημένη βάση αποτελεσμάτων και το κάθε έργο να αξιολογείται με δείκτες παρακολούθησης προσθετικότητας. Στην παράγραφο 20 αυτά. Για να επιτευχθεί η προσθετικότητα προφανώς έχει μεγάλη σημασία. Η διοίκηση, τα είπε ο κύριος Σάρβαμα, ο κύριος Συγητής, ε, διαφάνεια, απλοποίηση. Θεωρώ πως ο εισηγητής θα μπορούσε να είναι πιο σαφής εδώ πέρα γιατί ζητάει με ήπιους τόνους καλύτερη διοίκηση. Λέει στην παράγραφο 4 ότι θεωρούμε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια για να υπάρχει αποκαλύψη των πληροφοριών και των ε, λειτουργιών μέσω του πίνακα βαθμολογίας δικτών. Πρέπει να το πούμε πιο έντονα δεδομένων και των σχολείων που έκαναν οι συνάδελφοι και να επιμείνουμε στην ε, πραγματική διαφάνεια. Επίσης, στην παράγραφο που περιέλαβε ο συνάδελφος που ζητάει να οριστούν καλύτερα οι ευθύνες που αντιστοιχούν σε Κομισιόν και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, ειδικά όσον αφορά τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Και αυτό πρέπει να το πούμε πιο ξεκάθαρα και πιο έντονα ως Κοινοβούλιο. Μετά, για το θέμα των γεωγραφικών ανισορροπιών. Εγώ θεωρώ, σε αντίθεση με κάποιους από τους συναδέλφους και τον κύριο Σάρβαμα, ότι σωστά λέει ο εισηγητής ότι ήταν άνηση η κατανομή και η συνοχή και η βιωσιμότητα θα πρέπει να εξασφαλιστούν με μια ευρύτατη γεωγραφική διασπορά και πάλι εδώ πρέπει να πούμε κάτι πιο έντονο από το θα πρέπει να εξεταστεί και σωστά τονίζουμε ότι δεν θα πρέπει να, θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο επενδύσεις, όχι εκεί όπου δεν χρειάζονται. Αυτή είναι δε μία ιδεολειψία από αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι υποεκπροσωπούνται στο θέμα των επενδύσεων, αλλά τελικά ένας ε, βασικός δείκτης του εάν επιτυγχάνεται η προσθετικότητα είναι το εάν υπάρχει καλύτερη γεωγραφική κατανομή. Θεωρώ ότι κάποιοι συνάδελφοι έχουν κάποια πράγματα ήδη στο μυαλό τους και θεωρούν ότι το να πηγαίνουν στις χώρες ε, τις 13 τις λεγόμενες ε, θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος που σχετίζεται με παράνομες ή ύποπτες πρακτικές. Αλλά τα τελευταία πολλά χρόνια βλέπουμε μεγάλες επιχειρήσεις στις μεγάλες ε, βιομηχανικές χώρες, στις 15 παλιές όπως τις λέμε χώρες, με πολύ διεφθαρμένες ε, πρακτικές ε, και ε, σε πολλές περιπτώσεις ε, έχουν ε, κληθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και έχουν πληρώσει και πρόστιμα ή ποινές. Οπότε δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι όταν ζητάμε μεγαλύτερη γεωγραφική κατανομή μπαίνουμε σε χωράφια επικίνδυνα από την πλευρά της νομιμότητας. Θεωρώ και επαναλαμβάνω η γεωγραφική ισορροπία είναι ένα από τα κριτήρια επιτυχίας της προσθετικότητας. Έχω και κάποια στοιχεία. Οι 15 παλιές χώρες είναι 92% των υπογραφών και οι άλλες 13 χώρες το 8% των υπογραφών. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Τέλος ε, για την παράγραφο 27. Λέμε, επαναλαμβάνει τον ε, κέριο ρόλο του Κοινοβουλίου για την συμπληρωματικότητα και την προσθετικότητα. Αυτό. Συμφωνώ απολύτως και έχουμε πολύ ε, δρόμο ακόμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σημαντικές παρατηρήσεις αυτές. Επειδή αν κοιτάξει κανείς τον κανονισμό του προϋπολογισμού και τη σχέση μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του ΕΤΣΕ μπορεί να του έρθουν αμφιβολίες για το νόημα των μηχανισμών αυτών και να διερωτηθεί τι υπάρχει πίσω από όλο αυτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την γραμματότησή του. Είναι σημαντικό να την εξετάσουμε στα πλαίσια του ότι ετοιμάζουμε γνωμοδότηση για την Οικονομική Επιτροπή. Και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι τόσο η διαδικασία αλλά η ουσία, δηλαδή να καταλάβουμε κατά πόσον αυτό το χρηματοοικονομικό μέσο είναι το πιο δόκιμο για τους σκοπούς που έχουμε τάξει. Δηλαδή, αν βοηθά να ελκύσουμε επιπλέον επενδύσεις, να κινητοποιήσουμε ε, πόρους, ούτως ώστε να δοθεί όθηση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και να βοηθήσουμε ταυτόχρονα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εννοείται ότι συμφωνούμε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, αλλά βέβαια εδώ πρόκειται για το ότι θέλουμε να υπάρχει μια ανάλυση εις βάθος για το κατά πόσον αυτό το εργαλείο θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς που επιδιώκουμε ή αντίθετα για το κατά πόσον δεν θα αποδώσει σε σχέση με τους στόχους μας. Οπότε γι' αυτό θα ήθελα, εάν μπορούσε ο συγητής, να μας ε, δώσει μια σφαιρική εικόνα για το τι μπορούμε να βελτιώσουμε για όλη αυτή τη διαδρομή. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι είπε ότι είδα στο παράρτημα τι λέει για τα σχέδια αν μπορεί να μας τα, τα εξηγήσει για αυτά τα σχέδια τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να εγκριθούν αυτά τα σχέδια όσον αφορά την ουσία τους γιατί υπάρχει προσθέμενη αξία την οποία αποδίδουν. Νομίζω ότι τώρα έχουμε αυτή την ευκαιρία να ξαναδούμε με τι διαδικασία εγκρίνονται αυτά τα σχέδια. Υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή που ασχολείται ακριβώ με αυτό και αξιολογεί το περιεχόμενο ε, και το πόσο ωφελούν αυτά τα σχέδια. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση πάνω σε αυτό, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα και εγώ να μιλήσω. Στην γνωμοδότηση μου λείπει μια παραπομπή στη γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου για την επέκταση αυτή του ΕΤΣΕ. Ήταν τόσες σελίδες που ήταν μια εις βάθος ανάλυση που περιείχαν σημεία τα οποία θα μπορούσαμε ή μάλλον θα έπρεπε να επεξεργαστούμε και εμείς. Οπότε η ερώτηση προς τον εισηγητή είναι γιατί πουθενά δεν αναφέρεται η πρόθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχουμε την τάση ως κοινοβούλιο να ξοδεύουμε χρήματα και περισσότερα χρήματα είναι πάντα καλά. Αλλά το ελεγκτικό συνέδριο μας υποδεικνύει πως έχουμε πολλαπλασιασμό των αναγκών σε εγγυήσει και πως δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία. Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας του ΕΤΣΕ αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δηλαδή θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί το σημείο αυτό, αλλά να ασχοληθούμε επίσης με αυτό που είπε το ελεγκτικό συνέδριο, πως την αξιοποίηση και πως το ταμείο αυτό εντός της λειτουργίας του θα βελτιωθεί συγκεκριμένα. Αυτή η γνωμοδότηση είναι πολύ γενική, δεν είναι αρκετά συγκεκριμένη. Μπορούμε να τα παραμερίσουμε όλα αυτά λέγοντας ότι τα έχουμε ούτως ή άλλως. Εάν βάλουμε περισσότερα θα μπορέσουμε να επιτύχουμε περισσότερα, περισσότερο από ό,τι εάν λέμε γενικολογίες. Η συνάδελφος Άγια Λασένταρ ζήτησε τον λόγο, ευχαριστώ. Ακριβώς. Νιστάζουμε όλοι ακόμα. Δεν θα έλεγα ότι έχετε κακές προθέσεις. Σίγουρα είμαστε από την ίδια πλευρά. Δεν θέλω να αφισβητήσω κάτι τέτοιο. Η έκθεση αυτή, το ότι την εξετάζουμε, αυτό είναι θετικό. Βλέπουμε φυσικά και τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε, αυτό που επιτύχαμε ήδη, και επίσης μιλούμε γενικώ για τις διαδικασίες. Επίσης συμφωνώ με τον κύριο Κρίνσκι για την μη ισορροπημένη γεωγραφική κάλυψη. Αυτό είναι γεγονό. Και φυσικά τίθεται το ερώτημα για τα αίτια. Και πιστεύω πως αυτό οφείλεται ακριβώς το ότι στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη ενώ τις νέες χώρες φυσικά πως εκεί λείπει η ικανότητα προετοιμασίας έργων, με άλλα λόγια το capacity building. Πιστεύω πως αυτός είναι ένας τομέας τον οποίο μπορούμε να υποδείξουμε στην έκθεσή μας. Θέλουμε κάτι μεγάλο χωρίς να ξέρουμε αν μπορούμε να το κάνουμε. Αν μπορούμε να το πληρώσουμε και τότε λέμε πως το έτσι πρέπει να βοηθήσει. Αυτό σε τι θα καταλήξει με αυτή την προσέγγιση. Ακούμε και απόψεις σύμφωνα με τις οποίες το Ταμείο θα λαμβάνει χρηματοδότηση σύγκλησης, δηλαδή από τα νέα κράτη-μέλη, τότε οι ροές χρημάτων θα είναι μικρότερες Δηλαδή θα παίρναμε τη χρηματοδότηση αυτή από χώρε, οδηγώντα σε έλλειψη ικανοποίηση, αν και δεν είναι δικαιολογημένε όλε οι καταγγελίε, επειδή γνωρίζετε από ποια χώρα είμαι εγώ. Και τι κάνει η δική μας κυβέρνηση σε ευρωπαϊκές υποθέσεις. Γι' αυτό και είναι καλό εδώ να μην κατηγορούμε εσφαλμένα Κύριο Στάκουλα. Ήδη αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα με τα οποία συμφωνώ και από πλευρά μου θα ήθελα να συμπληρώσω το capacity building, ιδίω για τι χώρε που δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο και οι οποίες δεν κατανοούν ακόμα τη φύση του μηχανισμού αυτού. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ίνες, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια προς τον κύριο Τάκουλα. Νομίζω ότι τα πιο σημαντικά στοιχεία που έχουν πολιτική χρειά περιέχονται στο κείμενό του και από ό,τι βλέπω τα ίδια λένε και συνάδελφοι. Τώρα θέλω κάτι να σας πω όσον αφορά για το ελεκτικό συνέδριο. Να θυμηθούμε ότι για αυτό το θέμα Όπως και για το επόμενο, για την πρόταση παράτασης, ισχύω υπάρχει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων και αφορά αυτό κάποιο μέλος του Ελληνικού Συνεδρίου. Έχουμε εδώ εκπροσώπους του Ελληνικού Συνεδρίου και όλα αυτά ελπίζω να ξεκαθαριστούν στα πλαίσια του οργάνου αυτού. Ε, πρόκειται για κάποιον που ήταν επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό. Και μετά ε, μπερδευτήκαμε και με, το, με την ε, Τράπεζα Επενδύσεων. Τελικά διατυπώθηκαν κάποιες επικρίσεις ε, πάρα πολύ Οπότε δεν θα πρέπει να αδικούμε αυτή την υπόθεση που αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πόσο χρειάζονται επενδύσεις, πόσο χρειάζεται να αντιληφθούν πόροι από τον ιδιωτικό τομέα που λείπουνε είναι κάτι πολύ αναγκαίο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τις δημόσιες κρατικές επενδύσεις. Επίσης έχουμε και κάποια καλά μαντάτα ότι η ΕΤΕ πάντοτε ήταν συντηρητική η τράπεζα με την καλή έννοια. Και τώρα στο καινούριο ΕΦΣΥ και το λέω αυτό γιατί έχω αναλάβει δύο εκθέσεις για τις μεταφορές ήδη η ΕΤΕ είπε ότι θα πρέπει να συγκρατήσουμε τις ε, οικονομικές ανάγκες που αφορούν τις εγγύησεις. Πάνω από έναν χρόνο πέρασε για να προσπαθήσουμε να δούμε τι θα γίνει με τον κόμβο, με το ΙΡ, τι θα κάνουμε δηλαδή με τους ε, πόρους του ιδιωτικού τομέα. Οπότε έχουμε δεδομένες αυτές όλες τις κριτικές, βέβαια δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, αλλά θεωρώ ότι τελικά πρόκειται για υπόθεση πολύ θετική και μια τράπεζα σαν την ΕΤΕ που δεν χρειάζεται και τόσους πολλούς πόρους από τον προϋπολογισμό αφού τώρα ήρθανε και μειώσανε ε, τις εγγυήσεις κατά ένα σημαντικό ποσοστό ε, αυτό πιστεύω ότι σημαίνει πως το πρόγραμμα βαδίζει σε καλό δρόμο. Και οπότε όταν αρχίσει να λειτουργεί κανονικά όλα θα πάνε καλά. Βεβαίω και πρέπει να γίνει πιο ισόρροπη κατανομή ανά μέλος, μέλο ε, και θέλουν τα κρατημέλη να συμμετάσχουν πιο ε, ενεργά. Οπότε τώρα δείχνουμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάποια σχέδια, προγράμματα που ενέχουν κινδύνο, κινδύνους, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ. Για το θέμα της σύγκρουσης ε, συμφερόντων των μελών, από ότι η μόνη κατηγορία που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι ήταν ε, ειδικό και ήξερε ακριβώς ε, περί... και ήξερε περί τίνο μιλούσε γιατί είχε παρακολουθήσει το ζήτημα στο Συμβούλιο και ήταν εκπρόσωπος στο Συμβούλιο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχε και σύγκρουση συμφερόντων. Θεωρώ πω ε, καλά θα κάνουμε να λάβουμε υπόψη αυτές τις ε, παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, το οποίο ο θα το κάνει ούτω ή άλλως και θεωρώ ότι αυτό οφείλει πάρα πολύ γιατί η συστημική κριτική που έκαναν συνάδελφοι Λιμπερίτσκι και Πυρίνσκι πράγματι απευθύνεται και υπάρχει στο ΕΦΣΙ. Θεωρώ λοιπόν πως θα πρέπει να προσέξουμε αν δηλαδή δεν γίνεται να είναι έτσι τα πράγματα, θα πρέπει να έχει κάποιες βασικές αρχές το Εύση που θα το θωρακίσουν και πρέπει να, έχουμε κάποι, να πούμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Αν θέλουμε να επιτύχουμε μια γεωγραφική ισορροπία, κάτι το οποίο θέλουμε νομίζω όλοι, θα πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή στο Εύση προς αυτή την κατεύθυνση και να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις και να πω πως το ερώτημα γιατί έχουμε αύξηση μετά από ένα έτος ε, παραμένει αναπάντητο, αλλά θα λάβει τον λόγο η Κομισιόν. Λοιπόν, ο συνάδελφος ε, Σάρβαμα και μετά η κυρία Βαρτών από την ε, DG Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι και να ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο νομίζω έχει μεγάλη σημασία εδώ. Εμείς ως Επιτροπή Ελληνικού Προϋπολογισμού πρέπει να ζητήσουμε διαφάνεια. Αλλά τον... Ε, έχουμε τελικά διαφάνεια και πρόσβαση στα κριτήρια και στις ε, αποφάσεις ε, και στις ποιοτικέ πληροφορίες είναι το ένα. Αλλά το να προσπαθούμε μετά να αλλάξουμε τα κριτήρια είναι κάτι άλλο. Ε, θέλω να το πω λοιπόν αυτό εδώ. Θα ήθελα να ε, επανέλθουμε στο 2014-2015 όταν η Κομισιόν ε, επινόησε το σχέδιο αυτό. Και όπως υπόθηκε είμαστε ακόμα στις αρχικές φάσεις. Ο χρόνος πετάει όπως λένε. Περνάει πολύ γρήγορα. Αλλά είναι σαφές ταυτόχρονα ότι η πολιτική σημασία Καλά, ξέρω ότι θα το συζητήσουμε και στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Αλλά Η ίδια η ύπαρξη του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων έχει τόσο μεγάλη πολιτική σημασία έτσι ώστε σε αυτή την φάση δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα, τα βασικά στοιχεία του σχεδίου Γιονκέρα έχω την εντύπωση ότι ο Αντιπρόεδρος, ο Αρμόδιος Επίτροπος, λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει καν ότι υπάρχει αυτό το ταμείο και ότι απαιτείται διαφάνεια και επίσης αν κατάλαβα καλά τον κύριο Λιμπεράτσκι συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε όλα τα κράτη-μέλη. να έχουν καλύτερα επενδυτικά έργα. Στο ΔΕΕΦΣΙ υπάρχει κάποιο ζήτημα. Οι επαγγελματίες επιλέγουν τα έργα και έτσι πρέπει να συνεχίσει να έχει η κατάσταση. Και για να είμαι σαφής, εγώ δεν θέλω να αλλάξουμε τα βασικά κριτήρια επιλογής έργων ε, τα οποία θα είναι τα πιο βιώσιμα ανεξαρτήτως κράτους μέλους. Και υπ' αυτή την έννοια βεβαίω ε, είμαι υπέρ μια καλύτερη γεωγραφική ισορροπία, αλλά αυτό το οποίο προσπαθούσα να πω και αυτό το οποίο λέω είναι ότι πρέπει να γίνει μέσω βιώσιμων έργων. Και αν μπορούμε να βοηθήσουμε με τη διαφάνεια, με την επικοινωνία, με την πρόσβαση στα, κριτήρια, στα έργα. Και θεωρώ πως ε, πράγματι θα πρέπει τα κριτήρια επιλογής να είναι δημόσια και με διαφάνεια. Αυτός είναι ο δικός μας ρόλος ε, Λοιπόν, αυτό ήθελα να προσθέσω. Ε, κυρία Βαλτών, δεν ξέρω αν θα λάβετε τον λόγο για την εφαρμογή ή και για τα δύο. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ που δίνετε και στην Κομισιόν ε, την ευκαιρία να εκφραστούμε λίγο. Λοιπόν, μια που έχω την ε, δυνατότητα να μιλήσω φιλανδικά, θα το εκμεταλλευτώ. Να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Τάκουλα στα φιλανδικά. Κοιτάξτε, έχουμε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης του εισηγητή και άψω και προσεκτικά την σημερινή συζήτηση και θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια σημαντικά σημεία. Η γνωμοδότηση τονίζει πολλά ζητήματα που αναφέρθηκαν περιέχονται στην πρόταση της Κομισιόν για την επέκταση της πρότασης για το ΕΦΣΙ. Θα ήθελα να αναφέρω την αυξημένη διαφάνεια που ακούγοντας ε, τους ενδιαφερόμενους και άλλους εντός του Κοινοβουλίου περιλάβαμε χρησιμοποιήσαμε εντονότερες διατυπώσεις έτσι ώστε να εξηγούνται καλύτερα οι λόγοι επιλογής των έργων. Χρησιμοποιούμε και τον κατάλογο βαθμολογίας ε, και τις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων και αυτά μπήκαν στον κανονισμό υπάρχει ακριβώς καλύτερη πληροφόρηση για το πώς επιλέγονται τα έργα. Μια άλλη πτυχή είναι οπωσδήποτε η γεωγραφική κάλυψη και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το δούμε. Είτε κοιτάμε τα νούμερα ή κοιτάμε να δούμε αν η πλειοψηφία δεν είναι στις χώρες συνοχής αλλά αν δούμε την κατάσταση τα ποσά σε σχέση με το ΑΕΠ ε, θα έχουμε μια πιο ισορροπημένη νομίζω εικόνα. Αλλά αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και εδώ υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ακριβώς ε, ο κόμπος συμβουλών προς τους επενδυτές και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για να υπάρξει ακριβώς ε, η δυνατότητα αυτή στα κράτη-μέλη που δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία την δημιουργία δομών που θα επέτρεπαν στο ΕΦΣΙ να χρησιμοποιήσει έργα σε αυτές τις χώρες, αλλά το ΕΦΣΙ ακριβώ έχει σχεδιαστεί με βάση την ζήτηση. Ε, αλλά μπορούμε βεβαίως και να στηρίξουμε την ζήτηση σε κάποιες χώρες για να, για να κάνουμε καλές προτάσεις Θα κλείσω αναφέροντας ε, την ενισχυμένη προσθετικότητα. Η Κομισιόν το θεωρεί αυτό κάτι το πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, φορές, ε, πολλές φορές που έχουμε τονίσει ότι τα έργα πρέπει να είναι επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν προστιθέμενη αξία, να καλύπτουν κενά της αγοράς και κάναμε προτάσεις σε ποια κατεύθυνση θέμε να πάμε. Γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε διασυνοριακά έργα. λόγω της σημαντικής τους διάστασης για την Ένωση και καλό θα ήταν πράγματι το Ταμείο τελικά να στηρίξει την καινοτομία στην Ευρώπη παρέχοντας ε, χρηματοδότηση στους κίνδυνους. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο εισηγητής για να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τους συμβαδέλφους για τα καλά σχόλια για τα σημαντικά αυτά σχόλια. Δεν θα τα απαριθμίσω αλλά γενικά θα ήθελα να πω πως είμαι σίγουρος πως θα έχω την υποστήριξή σας κατά την περαιτέρω εκπόνηση της γνωμοδότησης αυτής. Ο συναδελφός Σάρβαμα ήδη ανέφερε σημαντικά ζητήματα όσον αφορά την γεωγραφική ισορροπία. Τι να πω. Και οι δυο μας είμαστε από μια μακρινή χώρα εσύ από το Ελσίνκι, εγώ από τη Λαπωνία, από το Βορρά. Και από ό,τι φαίνεται, μας λείπει η πίστη πως τέτοια έργα μπορούν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Πρέπει δηλαδή να διασφαλίσουμε πως θα λειτουργήσουν τα πάντα, αλλά φυσικά, όπως υπόθηκε πολλές φορές εδώ, πρέπει να θυμόμαστε πως η πολιτική σύγκλησης έχει το δικό της ρόλο και το ευσύ, το έτσε έχει έναν άλλο ρόλο δηλαδή τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις δραστηριότητες επενδύσεων στην προσέλκυσή του. Όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη, πρέπει να γεφυρώσουμε κατά κάποιον τρόπο το χάσμα που υφίσταται. Αλλά έχουμε ένα ταμείο, έχουμε τις δυνατότητες, γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε τη δυνατότητα αυτή. Επειδή θέλουμε να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία. Συνάδελφε Περίνσκι, αναφερθήκατε σε σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα ενσωματώσω στην εργασία μου. Έχετε δίκιο, υπάρχει μια καλή διατύπωση, το ζητούμενο είναι η καλύτερη διαχείριση και παρόμοια ζητήματα και πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να μπορέσουμε να εργαστούμε πιο αποδοτικά, με μεγαλύτερη διαφάνεια. Συνάδελφε Σαλαφράγκα, αυτά μόνο. Το πετύχατε ακριβώς μπήκατε στην ουσία. Έτσι πρέπει να γίνει και όχι με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να αναλύσουμε κατά πόσον με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους κάθε Και ό,τι και αν επιλέξουμε σε εθνικό επίπεδο, κατά την επιλογή των έργων. Στη Φιλανδία η μεγαλύτερη τράπεζα που είναι αρμόδια για τη διαδικασία επιλογής αυτής Μπορεί να διαρωτηθεί κανείς βέβαια πώς γίνεται η απόφαση. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά ως προς αυτό. Αλλά φυσικά πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό. Το ζητούμενο με το έτσι είναι να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία και με τον τρόπο αυτό να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και έτσι ώστε να επιτύχουμε ανάπτυξη, αυτό που προσπαθούμε εδώ και χρόνια. Φυσικά και εύχομαι από την πλευρά σας συγκεκριμένες προτάσεις. Όταν συνέταξα το πρώτο κείμενο για μας, και αυτό είναι μια διαδικασία μάθησης και εγώ μαθαίνω όλο και περισσότερα για τις λεπτομέρειες. Πέραν αυτού εδώ θύχθηκε και ένα σημαντικό ζήτημα όσον αφορά την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ίσως θα μπορούσαμε να επισέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό. Φυσικά και το συνέδριο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες. Οι θέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη με καλύτερο τρόπο. Αυτό το είπε και ο συνάδελφος Λιμπεράτσκι, μεταξύ άλλων. Λοιπόν, τα σημείωσα όλα και θα κάνω ό,τι καλύτερο για να βελτιώσω το κείμενο ως προς τα σημεία αυτά, αλλά όπως είπα, η εργασία του βουλευτή και η εργασία εδώ είναι ωραία κατά την έννοια ότι υπάρχουν πάντα πολλοί που βοηθούν. Θα προσπαθήσω να εκπονήσω ένα ισορροπημένο κείμενο το οποίο θα περιέχει όλες τις θέσεις που διατυπώθηκαν εδώ. Πιστεύω πως αυτό αρκεί αυτή τη στιγμή. Οπότε παραμένω με την παράκληση για περαιτέρω σχόλια. Η προθεσμία για τις τροπολογίες δεν λύγει σε λίγες ώρες. Έχουμε χρόνο. Ναι, στις 28 Μαρτίου, στις 2 το απόγευμα, έω τότε μπορούν να κατατεθούν τροπολογίες, οπότε περνούμε στο τέταρτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την γνωμοδότηση για την παράταση λειτουργία του ΕΤΣΕ. Συνάδελφε Τάκουλα, σε λίγο θα πάρετε τον λόγο για να παρουσιάσετε την γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ. Σκέφτηκα ίσως ε, να μιλήσω αγγλικά τι ακούστηκε αυτή η θεωρία συνωμοσία ότι και ο Πέτρη Σάρβαμα είναι από τη Φιλανδία και εκπρόσωπο τη ε, Κομισιόν και στο ελεγκτικό συνέδριο υπάρχει κάποιο Φιλανδό. Τέλο πάντων, δεν υπάρχει συνωμοσία. Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα τώρα. Μιλάμε για το μέλλον, μιλάμε για το λεγόμενο ΕΦΣΙ 2 και την ανανέωση του ΕΦΣΙ. Έχουμε την δυνατότητα να προτείνουμε βελτιώσεις στον μηχανισμό χρηματοδότησης. Όπως ξέρουμε, η Κομισιόν προτείνει στα 26 αυτά δισεκατομμύρια να προσθεθούν εγγυήσεις κεφαλαίου ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ε, και σκοπεύει η Κομισιόν να εξασφαλίσει 500 εκατομμύρια χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα για τις επενδύσεις αυτές. Συμφωνώ με αυτούς τους φιλόδοξους στόχους και είναι πολύ χρήσιμοι για την ευρωπαϊκή οικονομία. Πρότεινα κάποιες ε, τροπολογίες ε, και αλλαγές στην πρόταση της ε, Κομισιόν υπογράμισα την προσθεμένη αξία που έχουν οι επενδύσεις και πρότεινα επιπρόσθετη χρηματοδότηση για τον συμβουλευτικό Κόμπο Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία η χρηματοδότηση για τον κόμβο αυτόν για να υπάρχει ακριβώς μεγαλύτερη προσβασιμότητα και στις αεροκατοικημένες περιοχές όπως ανέφερα. Η σημασία της επικοινωνίας και της διαφάνειας είναι πάρα πολύ μεγάλη όταν μιλάμε για χρηματοδότηση. Ένα στοιχείο είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που έχουν μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για αυτό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και την δική σας πρόταση από αυτό. Σας ευχαριστώ. Πρέπει λοιπόν να ενσωματωθούν και οι άλλες παρατηρήσεις του Ενεκτικού Συνεδρίου. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητάει τον λόγο. Πέτρη Σάρβαμα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο, αλλά μια που είμαι ο Σκιώδης ε, εισηγητής του ΕΛΚ, θέλω να πω δύο λόγια. Ήδη αναφέρθηκε ότι η επέκταση του ΕΦΣΙ έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω ακριβώς των πολιτικών λόγων που βλέπουμε στην Ευρώπη. Γι' αυτό η Κομισιόν είχε αυτή την πρόταση. Γνωρίζοντας ότι θα υπάρχει κάποια κριτική αφού δεν υπήρχε αξιολόγηση αντικτύπου στο f 1 Όπως όμως αναφέρθηκε Ε, χρειάζονται αυτές οι επενδύσεις. Είναι τόσο μεγάλο το κενό, δεν έχουμε χρόνο, αλλά καλωσορίζουμε επίσης και την ε, επέκταση αυτή. Τώρα όσον αφορά την ουσία. Δεν ε, βλέπουμε εδώ πέρα ξεκάθαρες ημερομηνίες και κριτήρια για την διαφάνεια. Νομίζω είναι ενδιαφέρον και ε, θετική και η προσθήκη του εισηγητή στην ε, τροπολογία 1. Ενδιαφέρον το ότι ζητάει η βιοοικονομία να ληφθεί υπόψη Ε, δεδομένου του ότι πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος αναπτύσσεται ταχύτητα και όσον αφορά την καινοτομία και θα ήθελα να αναφέρω συγκεκριμένα την ε, ιδέα που ανέφερα ήδη. Δηλαδή, το πώς ε, θα μπορούσαμε με έξυπνο τρόπο να βελτιώσουμε την ε, γεωγραφική ανισορροπία. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα για την ε, τροπολογία 2 που αναφέρεται ρητός σε αυτό το ζήτημα και η ιδέα ότι πρέπει να γίνει μέσω της αυξημένης ε, χρήσης του Ευρωπαϊκού αυτού συμβουλευτικού κόμβου για υπάρχει ακριβώς καλύτερη γνώση σε όλα τα μέρη της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Αυτά για την ώρα. Πυρίνσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κάποιες πρόσθετες σκέψεις και από πλευράς μου. Σαφώς και πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας στην έκθεση αυτή του κυρίου Τάκουλα καθώς συζητούμε κάτι που θα καταλήξει σε μια λήψη απόφασης. Όσον αφορά την πρόκληση της υπέρβασης μιας αποτυχίας της αγοράς και μη βέλτιστης κατάστασης επενδύσεων που είναι η βασική πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η παράταση θα ήθελα να αναφερθώ στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση του εύρους των επενδύσεων. Και αυτό που επικροτώ σαφώς είναι αυτό της συμπερίληψης του ανθρωπίνου και του κοινωνικού κεφαλαίου και της σχετικής υποδομής. Επειδή σε συζητήσεις που συμμετείχα με διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις και ενώσεις από τον τομέα των κοινωνικών υποθέσεων αυτό ήταν ένα από τα κύρια ελλείμματα της δραστηριότητας του έτσε μέχρι στιγμής. Δηλαδή οι κοινωνικές προκλήσεις και η ανάγκη μεγαλύτερης δέσμευσης του έτσε για την υπέρβαση των προβλημάτων. Όσον αφορά τις περιφερειακές ανισορροπίες, συμφωνώ με αυτό που είπε ο εισηγητής πως πρέπει να υπάρχει μια <laughs> ενισχυμένη αποδοχή του ΕΤΣΕ σε λιγότερο ανεπτυγμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές. Καταλαβαίνουμε βέβαια τι εννοεί καθώς ε, έχει την καταγωγή από τη Λαπωνία της Φιλανδίας. Είναι κάτι το οποίο ανέκυψε και σε προηγούμενες συζητήσεις και πρέπει να αντιμετωπιστεί και συμφωνώ επίσης με αυτό που υπόθηκε πως αυτό πρέπει να γίνει μέσω αυξημένης χρήσης του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι ακόμα που είπε ο εισηγητής. Η βελτίωση των τεχνικών ικανοτήτων του κόμβου αλλά και η δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού του. Ο τίτλος της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλά για τεχνική βελτίωση του κόμβου. Ο εισηγητής δεν αναφέρθηκε στη δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού και πιστεύω πως αυτό, εάν είναι δικαιολογημένο, πρέπει να υποστηριχθεί δηλαδή όχι απλά να δώσουμε περισσότερα χρήματα, έτσι ώστε να συνεισφέρουμε ενεργά στον, στην γεωγραφική διαφοροποίηση, όπως το ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά τις προκλήσεις για την διακυβέρνηση, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον εισηγητή όσον αφορά το άρθρο 414 ότι η ειδική εστίαση στην προσθετικότητα κατά την βελτίωση των εγγύσεων θα πρέπει να δοθεί όχι μόνο όσον αφορά τα αυστηρά κριτήρια προσθετικότητας αλλά επίσης με τους στόχους της ενωσιακής πολιτικής. Και εδώ ο πίνακας βαθμολογίας για την αξιολόγηση των έργων πρέπει να γίνει δημόσιος. Συγγνώμη τώρα θα κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή. Λυπούμε, θα σας διακόψω. Παρακαλώ σηκωθείτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι δύσκολο να συνεχίσω μετά από ένα τέτοιο λεπτό σιγής καθώς πριν θυμάμαι που ήμασταν πριν από ένα χρόνο. Οι περισσότεροι από εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο. Ολοκληρώνοντας όμως και επανερχόμενος σε αυτό που είπε ο κύριος Σάρβαμα σχετικά με το έως πού μπορούμε να φτάσουμε και αν έχουμε κατά νου να αλλάξουμε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Τραπέζας Επενδύσεων. Δεν νομίζω πως αναφερόμαστε σε αυτό, αλλά στην βελτίωση των μέσων, των τρόπων λειτουργίας του Ταμείου, έτσι ώστε να επιτύχουμε στόχους σύμφωνα με τα βασικά κριτήρια το οποίο δεν αφισβητεί κανείς. Ότι πρέπει να γίνεται μια ορθή επιλογή και εφαρμογή. Το ζητούμενο είναι το εξή. Δεδομένων των κριτηρίων αυτών, όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, υπάρχει ανάγκη να ληφθούν υπόψη πολλής βάθος τα εργαλεία, οι προσεγγίσεις της διαχείρισης, οι πρακτικές που υπάρχουν για να επιτευχθούν τέτοιοι στόχοι. Αυτό πιστεύω πως πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Σαλαφράνικα, ο επόμενος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πάλι συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σύμφωνο με την πρότασή του να έχουμε θετική στάση όσον αφορά την ε, πρωτοβουλία της Επιτροπής, τόσο ώστε να διευρυνθούν ε, οι πρόθεσμίε η διάρκεια τέλος πάντων. Ε, πρόκειται για τις ε, βελτιώσεις παράταση λειτουργίας του Ταμείου, όπως και είπαμε και προηγουμένω για το προηγούμενο θέμα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ποιοι είναι στο Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έφτιαξε αυτό το Ταμείο η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπαμε ότι σε πρώτη φάση πετύχαμε αυτό που θέλουμε αν μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς να δούμε κατά πόσον με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ε, ανάγκες της χρηματοδότησης και της πρόσβασης στο ιδιωτικό κεφάλαιο που ζητάει η αγορά και στη συνέχεια επίσης να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ε, λειτουργία του Ταμείου. Καλύτερη γεωγραφική ισορροπία, περισσότερη διαφάνεια, και ο στόχος όμως του Ταμείου δεν είναι αυτός. Δεν είναι η διαφάνεια και η γεωγραφική ισορροπία. Ο στόχος είναι το να μπορούμε να έχουμε ένα ε, ε, σχέδιο ούτω ώστε να μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση, να βοηθήσουμε στο να δημιουργηθεί απασχόληση και να ε, μπορέσουμε επίσης να επιλύσουμε τα σοβαρά προβλήματα της οικονομίας μας μετά την κρίση. Άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πρώτα-πρώτα τους στόχους για τους οποίους θα βοηθήσει το Ταμείο και από την άλλη μεριά της συνθήκη λειτουργίας. Νομίζω ότι σε αυτή τη βάση θα πρέπει να προχωρήσουμε πρόεδρε, αλλιώς ε, ε, θα, θα επικρατήσει σύγχυση. Πρόεδρος. Η Βάλτονεν της ε, Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστώ για αυτή τη γνωμοδότηση τον εισηγητή. Θέλω Να σας πω τα εξής ολίγα. Βεβαίω και θα υπάρξει ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε και στον ε, τριμερή διάλογο που θα συζητήσουμε τις ε, τροπολογίες και είχα την ε, αίσθηση ότι πολλά από αυτά που ελέγχθησαν ενισχύουν την πρότασή μας γιατί είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος οπότε να μην επισέλθω στις λεπτομέρειες. Πάντως ακούγοντας τη συζήτηση θα ήθελα να σας πω τα εξής. Βεβαίως και θα πρέπει να έχετε διαπιστώσει ότι θα έχουμε μία σειρά από αξιολογήσεις του προγράμματος ε, για το ΕΦΣΕ. Επομένως, ευθύς εξ αρχής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαπίστωση ότι σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτό το περιβάλλον θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πορεία, θα πρέπει έτσι να τονωθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρώπη, αλλά ε, χρόνο παραχρόνο θα γίνεται αυτή η αξιολόγηση από τους ε, ε ανεξάρτητους ειδικού για το πώς πάνε τα πράγματα. Ήθελα να σας το πω αυτό γιατί σχολιάστηκε. Ζητήθηκαν τέλος πάντων περισσότερα στοιχεία για αυτό το σημείο. Α, αυτό, αυτό προς το παρόν. Οπότε και περιμένουμε να συνεργαστούμε και στη συνέχεια στα πλαίσια της νομοθετικής πρότασης. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ σημαντικό που να ενσωματώσουμε τις ιδέες του ελεγκτικού συνεδρίου στην γνωμοδότηση, επειδή είναι σημαντικό αυτό. Ο συγκητής στο τέλος. Παρακαλώ. Τάκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα όσα είπανε. Και εγώ προχωρώντας μαθαίνω. Πολύ μεστά τα σχολιά τους και θα τα λάβω υπόψη. Αυτά προς το παρόν. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε τελειώσαμε το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης και έχουμε το πρόβλημα ότι μας λείπουν οι επόμενοι εισηγητές. Τώρα έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο συναδελφός Τάραντ θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ για να παρουσιάσει την γνωμοδότησή του και τώρα το ζήτημα είναι θα μπορούσαν οι πράσινοι είναι κάποιος εδώ Ο κύριος Τάραντ έρχεται. Πότε θα φτάσει? Σε λίγα λεπτά ελπίζω. Έχει ήδη αργήσει 8 λεπτά. Κανονικά ήταν στις 10. Οπότε διακόπτω τη συνεδρίαση για 5 λεπτά. Λυπούμε γι' αυτό. wir nehmen unsere beratungen wieder auf. ich möchte ich möchte dem kollegen Tarant auch gleich das wort θα ήθελα να δώσω κατευθείαν το λόγο στον συνάδελφο Τάραντ για να μας παρουσιάσει την κρομοδότησή του. Κύριε Τάραντ, έχετε το λόγο. to present your, you have the floor to present your... Έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε την γνωμοδότησή σας για το Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη που άργησα, αλλά υπήρξε η λυπηρή επέτειος της τρομοκρατικής επίθεσης, οπότε δεν μπόρεσα να προσέλθω από τη συνηθισμένη είσοδο. Πολύ γρήγορα όσον αφορά τη γνωμοδότηση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης το οποίο αποτελεί τμήμα της δεσμής μέτρων μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης γι' αυτό και ίσως είναι πιο σημαντικό από τη συνήθως παράλληλα γίνεται η παράταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και την αναθεώρηση των χρηματοπιστωτικών κανονισμών. Γι' αυτό θα πρέπει να παραμείνουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας, αλλά κάποιες φορές είναι χρήσιμο να υπερβούμε τα όρια αυτά και να συζητήσουμε εδώ. Τι θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα σχόλια και την κριτική που εκφράστηκε από το ελεγκτικό συνεδρίο όσον αφορά τα διαφορά χρηματοπιστωτικά εργαλεία το ελεγκτικό συνέδριο δεν τα αμφισβητεί αλλά τονίζει πως δεν λειτουργούν σωστά και πως κάποιες βελτιώσεις θα μπορούσαν να γίνουν. Σχετικά με αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ό,τι φαίνεται δεν έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές. Δεύτερον, ανησυχώ πολύ για τον τρόπο χρηματοδότησης του ΕΤΒΑ με μετάβαση χρημάτων από αναπτυξιακά έργα προς επενδύσεις αυτό προλυαίνει το έδαφος για να εξασθενήσει την αναπτυξιακή μας πολιτική με έργα που είναι ενάντια σε αυτό που χρηματοδοτούμε. Αν λάβουμε υπόψη τις γραμμές του προϋπολογισμού σε σχέση με την ανάπτυξη. Τρίτον, το κύριο σημείο κριτικής επί του λεγόμενου σχεδίου Juncker είναι η έλλειψη προσθετικότητας. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο λάθος και πρέπει να μάθουμε από τις εμπειρίες που αποκτήσαμε. Περαιτέρω, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά τους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς για το ΕΤΦΑ και τα κονδύλια του ΕΤΣΕ κατά την απόψή μου πρέπει να εστιάσουμε σε τρία ζητήματα την, τον δημοκρατικό έλεγχο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτό είναι κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα επειδή πιστεύω πως το Κοινοβούλιο αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Δομής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη περισσότερο την άποψη του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο επίσης. Δε, δεύτερον, ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Τρίτον, ενίσχυση, βελτίωση των συνθήκων χρήση του ΕΤΒΑ για να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του Ελεκτικού Συνεδρίου και για να γίνονται σεβαστοί οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω πως η Επιτροπή μας Ελέγχου του προπολογισμού θα διασφαλίσει πως ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι αποδοτικός και αποτελεσματικός ως προς την επιτευξή των στόχων που συμφωνήσαμε και ότι θα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα που συνάδουν με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την επίτευξη συμβατότητας του ΕΤΒΑ με τους στόχους Υπάρχουν τροπολογίες όπως η τροπολογία 11, την οποία θα ήθελα να προσέξουν οι συναδελφοί μου. Σύμφωνα με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ατζέντα 2030. Αυτά είναι όλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η πρώτη είναι η κυρία συνάδελφος Σμιτ. Ευχαριστώ. Το FST είναι κάτι το πάρα πολύ λογικό γιατί στον αφρικανικό χώρο όπως γνωρίζουμε χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη για να υπάρξει ευημερία των ανθρώπων και να μείνουν εκεί στον τόπο τους. Όμως ε, μπορεί τελικά το ΕΦΣΙ να αντισταθμίσει ακριβώς ε, το φαινόμενο της ε, φτώχειας. Αυτά για τα θετικά. Αυτό το οποίο δεν με ικανοποιεί είναι τα πρακτικά της κοινή αυτής ε, συνεδρίασης ΑΦΕΤ ΔΕΒΕ και τα όπου λέμε πως αυτή είναι η κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρά το ότι αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι χώρες ε, τέρη και οι διεθνείς ψηφιακοί οργανισμοί μπορούν να ζητήσουν καθεστώς ε, παρατηρητή. Πώς ε, θα γίνει, ποιος θα αποφασίσει αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ή Και επίσης αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί πιθανώς μέσω μιας θέσης στην μόνιμη επιτροπή του EFST. Και μετά τίποτα άλλο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Η Κομισιόν ε, το ήθελε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μετά παίζει τον κύριο ρόλο και εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά. Οι πολιτικοί θα μείνουν ε, απ' έξω, αλλά και πάλι θα εγκρίνει ένα σωρό λεφτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε αυτή τη φορά να αναφερθούν αυτά τα πράγματα, αυτή η σκέψη που αναφέραμε. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην εγκρίνει απλώς ε, πράγματα τα οποία δεν ε, ελέγχει εις βάθος και είναι εκτός, θα πρέπει να είναι μέσα και κοντά για να ξέρει το τι Θα πρέπει λοιπόν να έχει έναν πιο έντονο ρόλο στο ταμείο αυτό. Για να περιοριστεί ίσως κάπως και η δυσπιστία κάποιων συναδέλφων. Γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά και είναι νομίζω αναγκαίο και ένα σωστό μέσο για να επιτύχουμε τους ε, στόχους που έχουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος τον λόγο. Ε, να πω πως ε, πράγματι ε, όσο απλώς εγκρίνουμε χάνουμε επιρροή. Έτσι. Δεν γίνεται αλλιώ. Και εγώ θέλω να σταματήσουμε να φτιάχνουμε οργανισμούς εκτός του προπολογισμού και έχουμε πάλι άλλο ένα τέτοιο μέσο και εγώ έχω πολλά και μεγάλα ερωτήματα για το αν ελέγχουμε πραγματικά όλα αυτά τα μέσα εκτός του δεν ξέρω κάποιον που να έχει όντω μία εικόνα της κατάστασης. Και βεβαίως ε, αυτό δεν είναι σωστό και για τους ε, φορολογούμενους. Είναι προβληματική η κατάσταση. Δηλαδή ακούγονται καλά αυτά σαν τίτλο στο Ταμείο ε, Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά αυτό δεν βοηθάει σε τίποτα. Λοιπόν για την Κομισιόν τώρα, κύριε Πλάνας από την DigiTevco και μετά θα ακούσουμε και τις άλλες διευθύνσεις Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, αλλά και όσους βοήθησαν για αυτό το κείμενο. Πρώτα, πρώτα να σας πω ότι πήγαμε σε αυτή την κοινή συνάντηση για την έκθεση και ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό που αποκόμισαμε μας άποψη για τους στόχους κλπ. Και, και από πλευράς ΔΕΒΕ επίσης. Οπότε θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τουλάχιστον κατά τη γνώμη μας είμαστε σε καλό δρόμο. Κάπως ε, δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται με την ε, μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση για το πρόγραμμα, αλλά να μην κολλήσουμε σε αυτό απλώς, να σας τονίσω. Ότι έχουμε τις παρατήσεις του Ελληνικού Συνεδρίου, αυτά που έχετε και στις τροπολογίες, και εμείς θέλαμε από την αρχή να εμπλακεί όπως ο λεκανισμός το ελληνικό συνέδριο στην υπόθεση του Πάντω Πάντως ε, οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις του Ελληνικού Συνεδρίου έχουν ληφθεί υπόψη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίω όσον αφορά την προσθετικότητα για το ότι κάθε φορά που εγκρίνεται κάποιο πρόγραμμα σχέδιο <clears throat> θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι υπάρχει προσθεμένη αξία. Αλλιώς δεν θα εγκρινόταν, δεν θα γινόταν το πρόγραμμα σχέδιο. Οπότε θέλω και πάλι να σας διαβιώσω ότι ο στόχος, ο στόχος του Ταμείου είναι να έχουμε επενδύσεις, ανάπτυξη και απασχόληση. Κάτι το οποίο είναι σύντονο με τους στόχους της ανάπτυξης για Αφρική και για την νέα χώρες. Επίσης έτσι αντιμετωπίζουμε τις αιτίες της μετανάστευσης. Πάντως ο στόχος ο σχετικός με τη φτώχεια δεν πρόκειται να φύγει. Όσον αφορά το δημοκρατικό έλεγχο και το ρόλο του Κοινοβουλίου, προτείναμε το Κοινοβούλιο να λάβει μέρος σε αυτή τη στατική επιτροπή που θα δώσει κατευθύνες γραμμές για το ε, πρόγραμμα αυτό στο οποίο εντάσσεται και το ΕΤΒΑ. Και όλα αυτά θα έχουν σχέση και με την πολιτική ανάπτυξη, αλλά και με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Επίσης, θέλουμε να σας ε, καθισχάσουμε ότι οι στόχοι σχετικοί με την φτώχεια πρόκειται να λυθούν υπόψη ή με την πλατφόρμα επένδυσης ή από ε, το εγγυητικό σκέλος. Α, κάτι τελευταίο, μια ματιά στον εγγονισμό και θα δείτε ότι έχουμε ε, προσέξει πάρα πολύ το να υπάρχει ετήσια έκθεση προς Κοινοβούλιο και Συμβούλιο και προς Ελληνικό Συνέδριο όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά, όσον αφορά τη διαχείριση και υπάρχει κάποια αξιολόγηση που προβλέπεται. Αφορά το σύνολο αυτής της πολιτικής έχουμε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Ε, γι' αυτό και η Επιτροπή ε, ασχολείται με τον κανονισμό και με το πρόγραμμα επενδύσεων. Πρόκειται για κοινή προσπάθεια από πολλές γενικές ε, διευθύνσεις, ανάπτυξης, εξωτερικής δράσης κλπ. Ακόμα και νομική υπηρεσία έχει εμπλακεί. Έχουμε εδώ δύο συναδέλφους από την ε, από τα χρηματοοικονομικά και από την εξωτερική δράση. Δεν ξέρω αν θέλουν το λόγο. Ευχαριστώ. Ίσως πρέπει να πείτε και πόσες ε, θέσεις θα ε, μειώσει η Κομισιόν αν πάει πάλι η δουλειά στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Λοιπόν, θέλει τώρα ο κύριος ε, Μάρτιν τον λόγο. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, καλημέρα. Ναι, η ερώτηση αυτή είναι από τις πιο δύσκολες όπως ε, φαντάζεστε πώς θα μετρήσουμε τις δουλειές που δημιουργούμε ή που καταστρέφονται ή την ποιότητα των θέσεων εργασίας ε, που δημιουργούνται. Είναι πολύ δύσκολο ερώτημα για να απαντήσουμε όταν αναπτύσσουμε ένα μέσο ε, στον τομέα της εξωτερικής δράσης. Όχι μόνο επειδή είναι μεγάλη πρόκληση εντός της Ένωσης, αλλά και εκτός της Ένωσης γιατί τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε σε κάθε μία από αυτές τις χώρες ε, δεν είναι τόσο αξιόπιστα όσο αυτά που έχουμε εντός της Ένωσης. Οπότε αν βασιζόμαστε σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία και τα μετράμε ε, κάθε χρόνο εφαρμογής του έργου, βλέπουμε ότι η ποιότητα των στατιστικών αυτών στοιχείων είναι πολύ αμφίβολη και τα νούμερα αυτά αλλάζουν την αντίληψη για την κατάσταση στην ίδια τη χώρα πολύ πιο ριζικά από οποιαδήποτε αλλαγή μπορούμε να επιφέρουμε εμείς. Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε, αλλά βεβαίως όπως είπε ο συνάδελφος είμαστε αποφασισμένοι να προσπαθήσουμε να βρούμε το καλύτερο πλαίσιο αναφοράς και αξιολόγησης και παρακολούθησης για να έχετε εσείς ε, και το Συμβούλιο και ο φορολογούμενος ε, την καλύτερη ποιότητα πληροφόρησης για το τι έχουμε επιτύχει. Θα ήθελα λοιπόν να συμπληρώσω αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι η αντίληψη που είναι τελείως λάθος. Ε, θεωρούμε εμείς ότι το EFSD θα πάρει λεφτά από τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης σε ένα μέσο το οποίο είναι μέσο αναπτυξιακών τραπεζών και άρα δεν είναι αναπτυξιακό ταμείο. Δεν είναι σωστή αυτή η προσέγγιση. Το σκεπτικό εδώ είναι ότι τα ταμεία τα κονδύλια με συγχωρείτε της ανάπτυξης δεν μπορούν να πάνε μέσω απλών ε, επιχορηγήσεων. Γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιούμε πολλούς ε, ε, διάβλους κατά το οποίο βεβαίω είναι θετικό γιατί έχουμε 40 χρόνια αναπτυξιακή συνεργασία και βλέπουμε ότι οι επιχορηγήσει είναι λίγε, πολύ περισσότερο σήμερα. Οπότε δεν είναι δυνατό να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε χρησιμοποιώντα μόνο επιχορηγήσει. Ε, γι' αυτό θεωρούμε ότι το μέσο αυτό είναι μια καλή εναλλακτική για την χρήση ε, απλά επιχορηγήσεων. Γιατί υπάρχει και η μόχλευση επί 10, επί 11 και η εφαρμογή βεβαίως θα μας πει τι γίνεται στην πραγματικότητα, αλλά η εμπειρία μας δείχνει ότι είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο, οπότε μπορούμε να μοχλεύσουμε πολύ περισσότερα χρήματα για υποδομές ε, που χρειάζονται, για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρειάζεται στις χώρες αυτές. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι το Στρατηγικό Συμβούλιο θα έχει ε, έναν παρατηρητή από το Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η δικιά μας η πρόταση. Και θεωρούμε ότι έτσι δεν ε, θα μπορέσετε μόνο να δείτε το τι θέλουμε να κάνουμε στο EFSD, στον πυλώνα 1, αλλά να παρακολουθείτε όλες τις πληροφορίες που θα δίνουμε στο Στρατηγικό Συμβούλιο για την τεχνική αρρωγή, για το επενδυτικό κλίμα στην κάθε χώρα, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά ε, θέματα και πτυχές που δεν εξετάζονται συχνά. Δηλαδή το ότι θέλουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, όχι μόνο στα όσα κάνουμε από πλευράς επενδύσεων, αλλά και όσον αφορά την επένδυση του επιχειρηματικού κλίματος, βελτίωση των αγορών, των μη τραπεζικών επενδύσεων στις χώρες αυτές κτλ. Οπότε έτσι θα βελτιωθεί η παρακολούθηση των όσων κάνουμε στις χώρες αυτές από πλευράς επενδύσεων και επιχειρηματικού κλίματος και είναι σημαντικό νομίζω να το τονίσουμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται τα χρήματα δεν ρέουν από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε διερωτώμε πόσα κονδύλια ακόμα θέλουμε να θεσπίσουμε. Κυρία συναδελφέ, κάντε να αφήσουμε την κυρία Ραϊμόντι. Παρακαλώ. Ένα στόχο των προγραμμάτων αυτών είναι η ανέβρεση επενδυτών. Οπότε η ερώτησή μου είναι γενική. Σύμφωνα με ποια κριτήρια επιλέγεται κάποιος ως επενδυτής. Εδώ στο Κοινοβούλιο μιλήσαμε για ξέπλυμα χρημάτων τα τελευταία, τις τελευταίες μέρες. Γνωρίζουμε ότι πολλές αγορές λαμβάνουν με τεράστια τόνωση από επενδυτές από την Κίνα. Η ερώτησή μου είναι υπάρχει ένας κατάλογος κριτηρίων για το ποιοι επενδυτές να μάνονται υπόψη ή οποιοδήποτε είναι καλοδεχόμενος που φέρει λεφτά. Εκούνιαν Όλεπς, παρακαλώ. Ο κύριος Μάρτινς ή ο κύριος Πλάνενσπερκ, ποιος αυτοθυσιάζεται. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα απλά να σας βεβαιώσω κάποια πράγματα οι περισσότερες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται γίνονται μέσω διαπιστευμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ευρωπαϊκών ή όχι, επενδυτικών τραπεζών με μεγάλη παράδοση. Επίσης με περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες. Θέλουμε να προχωρήσουμε, αλλά σίγουρα θα διασφαλίσουμε πως τίποτα από αυτά που υπονοούσατε θα πραγματοποιηθεί. Υπάρχει το άρθρο 20 του κανονισμού Εκεί γίνεται σαφής αναφορά για τις, στις δραστηριότητες και στην μη συνεργατική δικαιοδοσία και στη μη υποστήριξη δραστηριοτήτων που γίνονται για, από το οργανωμένο έγκλημα που ευνοούν τη διαφθορά και τις αρχές της Ένωσης. Έχουμε πλήρη συνείδηση των ανησυχιών που θέτεται και θα το λάβουμε σαφώς υπόψη κατά την εφαρμογή του προγράμματος. Ευχαριστώ. Ναι, ενημέρωση προς το οργανωμένο έγκλημα. Ναι, αυτό απαγορεύεται. Κυρία Ρεμόντι, να ζητήσω την τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Και εγώ να σας διαβεβαιώσω. Χθες έγινε αυτή η συνάντηση με τις τρεις επιτροπές. Και με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι οι συνάδελφοί σας στην Επιτροπή Ανάπτυξης ήταν την πρότασή μας ακριβώς όπως και εμείς ότι δηλαδή πρόκειται για ένα μέσο προς των στόχων της ε, βιώσιμης ανάπτυξης πρόκειται για μια μακρόπνοη προσέγγιση. Α, ας πούμε, μας είπαν για το διεπιστήμα για την Αφρική, το οποίο έχει ξεκινήσει τι αστριότητέ του, αλλά μιλάμε και για κάτι μακρόπνο. Και η κυρία Μογκερίνη, όπω γνωρίζετε, ενδιαφέρεται πάρα πολύ να δει ότι θα ανέβει ο από τα δί στα τρει όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη γιατί δεν αρκεί μέχρι σήμερα ανθρωπιστική βοήθεια οπότε και είπαμε ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε νέους τρόπους ούτως ώστε να κινητοποιήσουμε χρηματοοικονομικά μέσα για τη βιωσιμή ανάπτυξη. Οι στόχοι ε, ODA, οι στόχοι αυτή τη ανάπτυξη δεν αρκούν, άρα θα πρέπει να κινητοποιήσουμε και ιδιωτική χρηματοδότηση, ε, τοπική, χρήματα δηλαδή που ήδη υπάρχουν στην Αφρική, αλλά τα οποία εκραίουν προς την ε, Ευρώπη. Άρα, να μείνουν τα κεφάλαια αυτά στην Αφρική και να γίνουν παραγωγές επενδύσει και να δημιουργηθεί απασχόληση εκείνη που χρειάζονται οι νέοι στην Αφρική. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε βιώσιμη απασχόληση, αξιοπρεπή απασχόληση. Και έτσι θα αντιμετωπίσουμε και τις αιτίες της μετανάστευσης. αν έχουν προοπτικές και ελπίδα οι νέοι, αν μπορούν να ζήσουν ειρηνικά, έτσι πετυχαίνουμε τους στόχους που είχαμε. Ε, βέβαια, η περιορισμένη εγγύηση δεν αρκεί. Γι' αυτό και είπαμε να γίνει σφαιρική συνολική προσέγγιση. Δεν μιλούμε μόνο για μια μικρή προσέγγιση. Χρειαζόμαστε τεχνική αρρωγή και όχι μόνο για τα σχέδια αλλά να μπορέσουμε να πλαισιώσουμε τους νέους επιχειρηματίες, τις ΜΜΕ και να μπορέσουν να έχουν βιώσιμα προγράμματα. Πέρα πέρα συνέργεια και με τους στόχους του G20. Δεν αρκούν τα χρήματα. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερο μετεδικο κλίμα. Θα πρέπει να έχουμε μεταρρυθμίσεις καταπολέμηση της διαφθοράς. Δεν είναι επομένω μόνο το θέμα αυτών των χρημάτων. Το τι κάνουμε δηλαδή με το Ταμείο Ανάπτυξης, το EDF και να εστιάσουμε προσοχή μας στην απασχόληση. Γι' αυτό και έχουμε και τις αντιπροσωπείες μας. Όπου, επί τόπου, έχουν εικόνα του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χώρες αυτές. Κάποιοι από εσά δεν μαρτυρήθηκαν, αμφισβήτησαν το overview που έχουμε. Ένα ε, τώρα βλέπετε τι έχουμε πετύχει εκεί και τώρα με το ΕΡΒΑ. Εκεί στοχεύουμε απασχόληση και ελπίδα για τους νέους της Αφρικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά. Προσοχή Νάρκες. Επειδή επί χρόνια βλέπουμε τι γίνεται με τα χρήματα, τι συνέβη μέχρι στιγμής με τα χρήματα, φυσικά και βρισκόμαστε στο πλάι σας σε όλα αυτά τα θέματα και η έλλειψη αποτελεσμάτων είναι αυτό που μας απασχολεί εδώ και χρόνια. Επίσης η συνεχής αντικατάσταση των μηχανισμών μας. Οπότε έχουμε πάντα τα προβλήματα εκκίνησης ε, που επηρεάζουν τα αποτελέσματα που αποβαίνουν εις βάρος των αποτελεσμάτων και όταν τα κάνουμε όλα ξανακάνουμε κάτι καινούριο και στο τέλος πάντα ίδια ιστορία και ακούμε πάλι την ίδια ιστορία ευχαριστούμε για αυτήν ο εισηγητής για το τέλος χαίρομαι πολύ για όλη αυτή την επιβεβαίωση. Αλλά θα ήθελα να σας επιβεβαίωσω και εγώ πως οτιδήποτε αφαιρεί τον έλεγχο από το Κοινοβούλιο θα με βρει αντίπαλο μέχρι την τελευταία σταγόνα θέματός μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, θέλατε, όχι. Κύριε Πλάνας, παρακαλώ. Θα ήθελα απλά να βεβαιώσω τα μέλη του Κοινοβουλίου πως σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε κάποια εξουσία από το Κοινοβούλιο. Θεωρούμε πως πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια. Αλλάζουμε τους τρόπους, μπαίνουμε σε πιο επικίνδυνα μονοπάτια και ζητούμε την κατανόησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς κατανοούμε σχεδόν τα πάντα. Ευχαριστώ. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 28 Μαρτίου στις 2 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ που ασχοληθήκαμε τόσο έντονα με το σημείο αυτό. Περνούμε στα Δυτικά Βαλκάνια, στο σημείο 6 ενίσχυση διοικητικών ικανοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια μεταέλεγχος, εισηγητής ο Γιώαχιν Τσέλερ μόλις ήρθε από την Ανατολική Ασία από το Ελεκτικό συνούδριο ο συνάδελφος Φάζακας που έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσω με την ε, παρουσίαση της έκθεσής μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, στον κύριο Γιώργη Τσέλερ, τον εισηγητή, και προσωπικά σε εσά για αυτά τα οποία κάνατε, το ότι καταφέρατε τόσο σύντομα να μπει αυτή η έκθεση στη σημερινή διάταξη. Θα θυμόμαστε όλοι ότι μόλις πριν από έναν μήνα στις 13 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο συζητήσαμε τα δύο θέματα της έκθεσης για την Ουκρανία και αυτής εδώ της έκθεσης. Αλλά λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος για την Ουκρανία όπου είχαμε πάνω από εννέα παρεμβάσεις δεν μπορέσαμε να ασχοληθούμε με αυτήν την έκθεση. Γι' αυτό το θέμα ήταν το πότε θα μπορέσετε να βάλετε το σημείο αυτό ξανά στην ημερήσια διάταξη σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι ε, θα μπορέσει και η αντιπροσωπεία του Μαύρου Βουνίου να, να παρουσιάσει μέρος αυτής της έκθεσης. Και σας ευχαριστώ που μπήκε στην ε, ημερήσια διάταξη. Επίσης, να σας ευχαριστήσω για το ότι μου δίνετε με την παρουσίαση αυτή η ευκαιρία να σας παρουσιάσω την τελευταία μου έκθεση το Κύκνιο. Άσμα μου, όπως ξέρετε, η εντολή μου τελείωσε με τον ορισμό της ε, διαδόχου μου Ε, Indigo και έτσι θα μπορέσω σε λίγους μήνες να αποσυρθώ και μάλλον αυτή είναι η τελευταία μου ευκαιρία να παρουσιάσω μια έκθεση. Έχουμε δύο-τρεις εκθέσεις ακόμα. Ε, ελπίζω μπορεί να ξανάρθω. Και θα ήθελα επίσης να πω πως ε, βεβαίως δεν είναι σωστό ένας πατέρας να ξεχωρίζει τα παιδιά του, αλλά αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιδιά, γιατί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον ε, Σεπτέμβριο στο Βέλιγράδι είχα διάφορες ε, ευκαιρίες να εξετάσω το θέμα. Μετά λοιπόν από αυτή την εισαγωγή να περάσω στην ε, έκθεση αυτή. Το πρώτο ερώτημα είναι τι είναι ο μεταέλεγχος. Λοιπόν, σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε την δουλειά που έχουν κάνει άλλο, δηλαδή, άλλοι. Δηλαδή, ο μεταέλεγχος καλύπτει μια σειρά σημείων χρησιμοποιώντας τις ε, ειδικέ εκθέσεις ΕΚΑ, ε, τις εξολογήσεις της ε, Κομισιόν και τις ε, εκθέσεις ε, πρόοδου. Έχουμε λοιπόν αξιολογήσει 52 εθνικά έργα στα Δυτικά Βαλκάνια και τρία έργα πολλαπλών δικαιούχων εστιάζοντας ιδιαίτερα στα θέματα του κράτους δικαίου και της ε, μεταρρύθμισης δημοσίας διοίκησης. Επισκεφθήκαμε λοιπόν την Κομισιόν της Αντιπροσωπείας και διαφορές δομές στα Δυτικά Βαλκάνια το ελεγκτικό συνέδριο χρησιμοποίησε την έρεια ε, που έχει τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουμε συντάξει 7 ειδικέ εκθέσεις για τα Δυτικά Βαλκάνια, τα βλέπετε στην οθόνη σας και βλέπουμε ή έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε το τι είναι το έργο το μέσο, με συγχωρείτε, προενταξιακής βοήθειας. Βλέπετε εδώ ποια είναι η κατανομή για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων από το 2007 μέχρι το 2013. Βλέπετε ότι η Σερβία ήταν ο μεγαλύτερος δικαιούχος του προγράμματος ε, αυτού και πως ακόμα και περιφερειακά ε, προγράμματα έπαιρναν ένα 23% της χρηματοδότησης που πήγαινε σε μια περιφερειακή προσέγγιση που έχει μεγάλη σημασία σε αυτήν την περιοχή γιατί έτσι υπάρχει διασύνδεση, περιφερειακή συνεργασία, ενίσχυση των ε, διοικητικών ικανοτήτων, κυρίως μέσω της διαδικασίας ε, του Βερολίνου. Μέσω κάποιων εργαλείων όπως το, ταμείο, το Επενδυτικό Ταμείο Δυτικών Βαλκανίων, την ε, Τοπική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και το Περιφερειακό Συμβουλίο Συνεργασίας. Γιατί λοιπόν έχει τόση σημασία το πρόταξιακό αυτό μέσο για τα Δυτικά Βαλκανία. Ε, δεδομένη της ε, σύγκρουση, ε, βλέπουμε πως υπάρχει οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά και το μέσο αυτό το προενταξιακό ακριβώς είναι το μόνο το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα της χαμηλής διοικητικής ικανότητας στη δημοσιοδιοίκηση την επιβολή του νόμου και στην δικαιοσύνη και στην διασύνδεση των χωρών αυτών και των χωρών που συνορεύουν με την Ένωση. Ποιε ερωτήσει κάναμε λοιπόν στην ειδική μα έκθεση. Η πρώτη ερώτηση είναι εάν η Κομισιόν διαχειρίστηκε καλά το μέσο αυτό στα Δυτικά Βαλκάνια και κατόπιν η δεύτερη ερώτηση εάν η αν το μέσο ενίσχυσε την διοικητική ικανότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Η πρώτη ερώτηση και πάλι. Αν διαχειρίστηκε καλά η Κομισιόν το μέσο. Βρήκαμε ότι η Κομισιόν δεν έθεσε πάντα συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, δεν εφάρμοσε συστηματικά αυστηρούς όρους και δεν τους παρακολούθησε, αλλά ήταν αποτελεσματική στην παρακολούθηση και αξιολόγηση και έπαιξε έναν θετικό ρόλο στο συντονισμό δωρητών στο επίπεδο των δικαιούχων είδαμε ότι οι κυβερνήσεις Αλβανίας, Βοσνίας, Ερζεγοβίνης και Κωσφοπεδίου είχαν μεγάλες ελλείψεις όσον αφορά τις αξιολογήσεις του κράτους Η απορρόφηση του μέσου εμποδίστηκε σε γενικές γραμμές από τη χαμηλή διοικητική ικανότητα και το Μαυροβούνιο και η Σερβία ήταν αποτελεσματικές στην ε, συνεργασία των δωρητών άλλες χώρες λιγότερο. Ε, έχουμε λοιπόν και κάποιες συστάσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι στο δεύτερο ε, μέσο με προτεραιότητες που θα έχουν μία σειρά καθώς και μετρήσιμους στόχους. Δεύτερον, να υπάρξει μία έμεση διαχείριση και επιλογή, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και την πολιτική ευαισθησία των έργων να υπάρχει αίρεσιμότητα σε όλα τα επίπεδα, να γίνεται συστηματική παρακολούθηση ευαίσθητων προγραμμάτων και έργων και εξωτερικές αξιολογήσεις σε τομείς προτεραιότητας. Το δεύτερο ερώτημα ήταν εάν το μέσο αυτό ενίσχυσε την διοικητική ικανότητα στα Δυτικά Βαλκανία για το κράτος δικαίου. Επειδή οι δικαιούχοι δεν είχαν αρκετό προσωπικό και στελέχωση, ούτε συντονισμό και ούτε πολιτική βούληση για μεταρρύθμιση των θεσμών, τα αποτελέσματα εν μέρη μόνο μπορούν να θεωρηθούν βιώσιμα και μόνιμα. Λίγη χρηματοδότηση πήγε σε συγκεκριμένους τομείς του κλάτους δικαίου, π.χ. την ε, εισαγγελία, την καταπολέμηση διαφθοράς ε, και του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης λοιπόν και η περιφερειακή συνεργασία. Υπήρχαν βιώσιμα αποτελέσματα σε πολλά έργα, αλλά ε, το μέσο μπορούσε να ενθαρρύνει τους δικαιούχους να τα χρησιμοποιήσουν για να διδαχτούν και άλλα κομμάτια της ε, δημόσιας διοίκησης. Το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας δεν είχε κάποια σημαντικό αντίκτυπο, αλλά όσον αφορά την Περιφερειακή Σχολή δημόσια Διοίκησης είναι πολύ νωρί ακόμα για να κρίνουμε την αποτελεσματικότητά τη Οι συστάσει μας για το θέμα αυτό είναι οι δικαιούχοι να εμπλακούν για να υπάρξει ακριβώ ένα πιστικό αποτέλεσμα όσον αφορά την διερεύνηση και δίωξη και καταδίκη της διαφθοράς υψηλού επίπεδου. Αυτό πρέπει να φανεί και στη μελλοντική χρηματοδότηση και στις άλλες πηγές ε, ευρωπαϊκής ε, χρηματοδότησης. Θα πρέπει να στοχεύουμε επίση καλύτερα τους πόρους σε συγκεκριμένους ε, τομείς του κράτους δικαίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και της ελευθερίας των ΜΜΕ. Και τέλος, αυτό βεβαίως το συζήτησα και με τον κύριο Γιώργη Μιτσέλερ, ότι πρέπει να στηριχθεί η περιφερειακή συνεργασία και το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας και η Περιφερειακή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ε, να έχουν μετρήσιμα και βιώσιμα αποτελέσματα επί το που είμαστε πεπισμένοι ότι η περιοχή αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ε, ως έξι μεμονωμένες υποψήφιες χώρες πρέπει να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση έτσι ώστε όλη αυτή η περιοχή να αναπτυχθεί για να ενταχθεί κάποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά για την έκθεσή μου. Χαιρόμαστε που α, ε, δημοσιεύτηκε και ε, βεβαίως υπήρχε και συνεργασία με Πελεγράδη και Σεράγιβο και σε στενή συνεργασία με την Κομισιόν Ελήθησαν υπόψη οι συστάσεις μας και η Κομισιόν ε, συμφώνησε μαζί, του, μαζί μας και αναμένουμε βεβαίως και την επανεξέταση εν καιρό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα έκθεση. Συστήνω να τη διαβάσετε επειδή φυσικά θα ασχοληθούμε με τη Σερβία και την περιοχή, θα ταξιδέψουμε εκεί το καλοκαίρι και θα κοιτάξουμε κάποια πράγματα για το και η έκθεση αυτή είναι μια πολύ καλή προετοιμασία. Ο συγκητής έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σόβετ Σάρακας και τις, τους συνεργάτες του για τη μεταέκθεση αυτή για την κατάσταση της προανεπτυξιακής βοήθειας της προενταξιακής βοήθειας πρόκειται για ένα γενικό απολογισμό αυτού που έγινε με τη χρηματοδότηση από την Ένωση στα κράτη αυτά. Επίσης είναι μια σύνοψη των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων για την κατηγοριοποίηση και εκτίμηση της κατάστασης. Μια τιτάνια εργασία, ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και πιστεύω πως τους επόμενους μήνες θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε πολύ καλά μαζί σας κύριε Φάσακας. Είμαι πεπισμένος πως αυτό θα πάει καλά. Τι απομένει να πω. Μετά την παύση της ύπαρξης της Ιουγκοσλαβίας στις αρχές της δεκαετίας του 90 και από τη διαδικασία διάλυσης αυτή προέκυψαν τα κράτη διάδοχη της Ιουγκοσλαβίας τα οποία είχαν μια δύσκολη διαδικασία, επώδυνη διαδικασία μπροστά τους, με εμφύλους πολέμους, με πολλά θύματα και μεγάλες τεράστιες ηλικές ζημίες. Στη συνέχεια, από τη διαδικασία σταθεροποίησης τα επιμέρους κράτη προσπάθησαν να αναπτύξουν τις κρατικές τους λειτουργίες το οποίο πέτυχε σε πολύ διαφορετικό βαθμό ενώ υπήρξε ένα κράτος, η Στοβενία, το οποίο εκπλήρωσε πολύ γρήγορα τα κριτήρια για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα στην Ευρωζώνη. Η Κροατία μπόρεσε να ακολουθήσω. Η κατάσταση στα υπόλοιπα κράτη της πρώην Ιγκοσλαβίας και πέραν αυτού στην Αλβανία που μας ενδιαφέρει εμάς είναι εντελώς διαφορετική. Εδώ η Κομισιόν κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες επένδυσε πολλά χρήματα και πολύ προσωπικό για να βοηθήσει τα κράτη αυτά να ορθοποδήσουν, να προωθήσει το κράτος δικαίου και την καλή διακυβέρνηση. και να δώσει στους πολίτες των χωρών αυτών τη συνείδηση πως η Ευρώπη δεν θα τους αφήσει μόνους τους αλλά αν κοιτάξουμε την κατάσταση στα επιμέρους κράτη πρέπει να διαπιστώσουμε πως ένα από τα κράτη αυτά δεν αναγνωρίζεται από όλα τα υπόλοιπα είναι το κοσυφοπέδιο. Επίσης όσον αφορά την πρώην Δημοκρατία της Δημοκρατίας υπάρχει το, η αντιδικία σχετικά με το όνομα δηλαδή πέρα, συν της άλλης έχουμε και πολιτικές δυσκολίες ως εμπόδια. Και επίσης διαπιστώνουμε πως πολλοί πολίτες έχουν χάσει τον ενθουσιασμό για την Ευρώπη. Το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε τρίτα κράτη εκ των έξω να ασκήσουν επιρροή εκεί. Παράδειγμα η Ρωσία, αλλά επίσης η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία τα κράτη αυτά θα μπορούσαμε να ονομάσουμε παραδειγματικά καθώς προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή στα κράτη αυτά. Αυτό φυσικά δεν διευκολύνει τα πράγματα καθώς τα κράτη αυτά και στο εσωτερικό τους είναι καθάλλου αποσταθερά, δεν διαθέτουν σταθερή διοίκηση, έχουν υπέρμετρες γραφειοκρατικές προδιαγραφές Έχουμε μια αμφίβολη διοικητική αποτελεσματικότητα. Μετά από εκλογές έχουμε μια μεγάλη αλλαγή πολιτικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού, το οποίο δυσχεραίνει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκεί. Γι' αυτό και η επιρροή αυτή είναι ένας πολιτικός στόχος τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε την αίσθηση στα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και κυρίως τους πολίτες που θα πρέπει να ανήκουν στην Ευρώπη. Αλλά πιστεύω πως θα χρειαστούμε πολύ περισσότερο από ό,τι σκεφτόμασταν στην αρχή μέχρι τα κράτη αυτά να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούν, να είναι όριμα προς ένταξη σύμφωνα με τα κριτήρια. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου δίνει πολύ καλές αποδείξεις σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει με τις οποίες συμφωνώ ως εισηγητής και πιστεύω πως εδώ δεν ζητείται μόνο το έργο της Κομισιόν κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων αλλά και τα κράτη-μέλη και η εξωτερική υπηρεσία θα πρέπει να προσέξει τα κράτη αυτά αν θέλουν να λαμβάνουν από εμάς βοήθεια ε, να πληρούν τις προϋποθέσεις που συνδέονται με την βοήθεια αυτή, δηλαδή την καταπολέμηση της διαφοράς, την διατήρηση καλής διακυβέρνησης και τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου, όπως και ο σεβασμός των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό πιστεύω πως θα, πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί θεμέλιο για την χορήγηση βοήθειας. Αυτό που μπορούμε να διαπιστώσουμε και αυτό που ακούμε από πολλά από τα κράτη αυτά είναι πως οι πολίτες δεν γνωρίζουν καν πως με πάρα πολλά χρήματα και προσωπικό βοηθούμε τα κράτη αυτά στη διαδρομή τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί απομένουν πολλά που πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε την ορατότητα των, της βοήθειάς μας το οποίο φυσικά είναι ζήτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά φυσικά και των εκεί κυβερνήσεων και των υπευθύνων στα κράτη τα ίδια. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε αναγνωρίσιμοι. Πως δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε πάρα πολύ τα κράτη αυτά στην πορεία τους και συνεχίζει να βοηθά, το οποίο θα κάνει και στο μέλλον πιστεύω. Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, επειδή όποιος παίρνει κάτι πρέπει να δίνει επίσης και εκεί πιστεύω πως απομένουν πολλά που πρέπει να γίνουν από πλευρά των πολιτικά ηθινόντων στα κράτη αυτά το οποίο και παρουσιάσαμε στην έκθεσή μας. Πιστεύω λοιπόν πως όπως είπε και η Πρόεδρος θα συνεχίσουμε να κοιτάμε πώς προχωρούν τα πράγματα εκεί. Δεν θέλουμε να χάσουμε σε καμία περίπτωση τα κράτη αυτά, αλλά επίσης και αυτό χρειάζεται η βούληση των κρατών αυτών. Πως αυτό που λένε πως θέλουν να προχωρήσουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνουν όντως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω υπάρχει πολύ πάθος εδώ, τόσο από το ελεγκτικό συνέδριο όσο και στην Επιτροπή αυτή, επειδή μπορούμε να κρίνουμε τα προβλήματα αυτά, έχουμε πάει τακτικά στο κοσυφοπέδιο, θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες σε όλα τα ασχοληθήκαμε με όλα τα κράτη, δώσαμε την αιγίδα μας σε όλα τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και τα κονδύλια που υπάρχουν για την περιφερειακή συνεργασία στην πρώην Γουσταβία βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ροή των κονδυλίων αυτών ή τουλάχιστον όχι όσο θα έπρεπε. Αλλά είναι ένα πρώτο βήμα για μια συνεργασία στην περιοχή, δηλαδή μια νομισματική ένωση, μια οικονομική ένωση, μια τελωνιακή ένωση κάποιου είδους επειδή αν ταξιδεύει κανεί στις χώρες της πρώην Ιουγκοσταβίας βρίσκεται αντιμέτωπος με καταστάσεις δηλαδή βλέπουμε τη διακοπή ροών κυκλοφορίας εμπορευμάτων στα σύνορα και είναι πολύ λυπηρό πως όλες οι πρωτοβουλίε που προβλέψαμε δεν ήταν επιτυχής. Ίσως η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να πει κάτι σχετικά με τα, τη χρηματοδότηση της περιφερειακής συνεργασίας. Τώρα δεν έχω κάποιον στον κατάλογο των ομιλητών που θα ήθελε να πει κάτι για το ζήτημα αυτό. Έτσι δεν είναι. Οπότε το επιβεβαιώνω, οπότε δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διτζινίερ, ο κύριος Γιούγκ, ανώτερος ειδήμων, σύμβολος του Διευθυντή. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ. Και επίση χαίρομαι που θεωρείται τόσο θετική συμβολή. Προσπάθεια με τις δύο εκθέσεις που είναι και δύο πάρα πολύ καλά ε, ε πάρα πολύ προσεκτικά διατυπωμένες και πρόκειται να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις επί τη βάση των όσων συστήνουν οι εκθέσεις. Κάτι ε, τα σημεία έχουν επισημανθεί, σαφώς. Ε, ελπίζω όμως ότι δεν θα πρέπει να ξεχνούμε πως ε, έχουμε μπορέσει να κάνουμε την διαφορά όσον αφορά την υποστήριξη από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περίοδο που προηγήθηκε ήταν δύσκολη έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα και καλές επιδόσεις στη διαδρομή. Παρά το ότι η πολιτική συγκυρία ήταν πάρα πολύ δύσκολη στις περιφέρειες γιατί είχαμε τις πληγές από τους πολέμους γιατί βέβαια οι ένοπλες συγκρούσεις συνεχίζονται στο μυαλό των ανθρώπων. Άρα δραματική αυτή η περίοδος και είχαμε την ε, χρηματοοικονομική κρίση του 2008 που χτύπησε τα Δυτικά Βαλκάνια σε μεγάλο βαθμό και μιλάμε για το 20% του πληθυσμού που έφυγε, μετανάστευσε από την ε, περιοχή. Οι δε οικονομικοί είναι πάρα πολύ χλωμοί όσον αφορά την ε, ανεργία και να των νέων γύρω Οπότε όσον αφορά τώρα την ε, εξέλιξη έχουμε αυτά τα δύο νομοθετήματα που οποία υπόψη και τις συστάσεις τους επίσης θα υπόψη και βέβαια θέλουμε από στατικής πλευράς να δούμε πώς θα επικεντρωθούμε σε κάποιους στρατηγικούς ε, κλάδους και να έχουμε κάποιο είδους μεταρρυθμίσεις ε, μεσοπρόθεσμες θα συμβάλλει γι' αυτό. Και να κινηθούμε στα πλαίσια και των ε, εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων για αυτούς τους κλάδους προτεραιότητας. Και θα γίνει στροφή σε σχέση με το τι κάνουμε στο παρελθόν. Θα επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα. Αυτό το πλαίσιο από τη βάση των ε, επιδόσεων, οι σχετικοί δείκτες και αυτοί και επίσης εποπτεία και παρακολούθηση και έλεγχος. Επίσης θα πρέπει να δούμε το, το πώς θα υλοποιηθούν αυτό που έχουν αποφασίσει για, για την αρρωγή και για τη βοήθεια, πώς θα αλλάξουν οι λεπτομέρειες. Έχουμε τώρα περισσότερα εργαλεία επίσης τώρα. Και έχουμε τους τομιακούς προπολογισμού Αλλά επίση θα υπάρχει τώρα αυτή η έμεση διαχείριση όσον αφορά του πόρου. Αυτό γίνεται από τι ίδιε τι χώρε, τι χώρε μέλη. Και είπαμε ότι τώρα θέλουμε να είμαστε ε, πιο προσεκτικοί, πιο ακριβεί στι ε, ενεργέ μα. Οπότε γι' αυτό και περικόψαμε του ε, πόρου που διαχειρίζονται οι ίδιε οι χώρε σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε τώρα πιο αυστηρέ προποθέσει, ούτω ώστε να υπάρξει πιο στιβαρή δέσμευση και βιωσιμότητα από πολιτική πλευρά. Οπότε, σε δύο χθε τι χώρε, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, είχαμε εντυπωσιακή μείωση της χρηματοδότηση. Βέβαια, την άλλη μεριά, όσο λιγότερη χρηματοδότηση έχει τόσο λιγότερα κάνει. Αυτό είναι τιμωρητικό κάπω. Αλλά θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να είμαστε προσεκτικοί στο πώς κινούμεθα. Οπότε έχουμε τα κίνητρα για περισσότερα αποτελέσματα. Έχουμε αυτή την αμοιβή. Το 13 θεσπίστηκε αυτό, ούτως ώστε να ανταμείψουμε κοινές τις χώρες που μπόρεσαν να προοδεύσουν σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις τους. Και όσον αφορά το ποσοστό της χρηματοδότησης στο παρελθόν. Επίση, ο προγραμματισμό τώρα είναι πιο σφιχτό σε σχέση με δράσει, με ε, σχέδια, προγράμματα για την υλοποίηση και δώσαμε βάρο περισσότερο στο θέμα τη οριμότητα και του χρονοδιαγράμματος για τις δράσεις. Υπάρχει πολιτικός διάλογος, υπάρχει μόχλευση, σύμφωνα με τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και αυτό θεωρούμε ότι είναι κίνητρο οι δικαιούχοι να προβούν σε μεταρρυθμίσεις, να υπάρχει η πολιτική τους δέσμευση και έτσι από πλευρά στήριξη να υπάρχει περισσότερη αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα. Θα συνεχίσουμε επομένω να ε, πιέζουμε για περισσότερη καταπολέμηση της διαφθορά και του οργανωμένου κλίματος. Αυτό βέβαια προποθέτει πολιτική δέσμευση από πλευρά ε, των αργών και απαιτεί και χρόνο. Επομένω θα προσφέρουν περισσότερο τα οικονομικά για τη διαχείρισή τους. Αυτό είναι θέμα που μα απασχολεί στα σοβαρά. οι ίδιες οι χώρες να διαχειριστούν τα δημοσιονομικά τους. Αυτή είναι η πρόκληση. Να γίνει όσο περισσότερο γίνεται καλύτερη η αξιολόγηση στο ιστορικό της χώρας. Η αξιοποίηση, συγγνώμη, των κοινωνικών κεφαλαίων και πόρων. Άρα θα αντίρρουμε τις προσπαθίες μας θα προσέξουμε και στο, στο 2 τη χρηματοδότηση Μεταρρυθμίσει επομένω οικονομική διακυβέρνηση, κράτος δικαίου. Οπότε για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων πρόκειται να δώσουμε του πόρου όσο χρειάζεται. Άπαξ Όμω και κυβερνήσει κυβερνήσεις προτίθενται να ασχοληθούν, να εμπλακούν με αξιόπιστο τρόπο για τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Εν κατακλείδη, θα συνεχίσουμε τη βοήθεια προς τα Δυτικά Βαλκάνια και προς το λαό τους. Και με τον πολιτικό διάλογο και με την χρηματοοικονομική βοήθεια, ούτως ώστε να φτάσουν τα ενωσιακά πρότυπα. Έτσι θα προετοιμαστούν αυτές οι χώρες για να γίνουν πλήρη μέλη της Ένωσης. Αναφέρθηκε σε αυτή η περιφερειακή προσέγγιση. Όντως. Αυτό όλο ένα και πιο σημαντικό γίνεται στο πολιτικό μας θεματολόγιο. Α, και την προηγούμενη εβδομάδα. Για πρώτη φορά. Από την εποχή του πολέμου είχαμε τους ε, υπουργούς των έξι χωρών τους πρωθυπουργού μάλλον που συναντήθηκαν στο Σαράγεβο για να συζητήσουν τι προτεραιότητες υπάρχουν, πώ μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα και ποιο θα είναι το αντικείμενο τη συνεργασία του. Υπάρχει βέβαια το, διαδικασία του Βερολίνου, η, το θεματολόγιο τη συνδεσιμότητα. Νομίζω ότι έχουμε δει πόσο σημαντική υπόθεση είναι η εμπλοκή και η δέσμευση που σταθερά ακολουθεί για τα Δυτικά Βαλκάνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επίση και τα συμπράσματα του τελευταίου Συμβουλίου. Κατατείνουν στο ίδιο. Ε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ενιαίος οικονομικός χώρος. Ενιαίος χώρος και οικονομικά Επομένω, γι' αυτό και συνεργαζόμαστε με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για να βρούμε μια προσέγγιση που θα οδηγήσει στην κοινή αγορά με βάση την οικονομία και τις ε, ελευθερίες. Να καταστρώσουμε σχέδιο δράσης με ορίζοντα το 2020. Να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε, τι πρέπει να πετύχουμε, τι, τι, τι δράσεις χρειάζονται και έτσι να οδηγηθούμε στο Συμβούλιο Κορυφής της 12 η Ιουλίου στην Τεργέστη της Ιταλίας όπου θα συνέλθουν οι χώρες οι πρωθυπουργοί των κρατών και να δούμε πώς θα γίνει αυτή η οικονομική διασύνδεση ή διασυνδεσιμότητα. Τώρα όσον αφορά την ε, προβολή ε, σε σχέση με το τι κάνει η Ένωση για να ε, υποστήριξη αυτές τις χώρες, θα πρέπει πάνω σε αυτό να προχωρήσουμε περισσότερο. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους προβολή. Τα συζητάμε και προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Να υπάρχει αυτή η προβολή σαν προτεραιότητα. Να καταπονιμήσουμε την παραπληροφόρηση. Για τα ψέματα, για το τι γίνεται που τα κυκλοφορούν κάποιοι που έχουν αντίθετα συμφέροντα. Έχουν συμφέροντα εντός και εκτός του ίδιου των χωρών. Ένα ε, είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά χρειάζεται αυτή η προβολή της δραστηριότητάς μας. Είναι βέβαια και θέμα υπομονής όσον αφορά αυτή τη διασύνδεση των οικονομιών. Για μεταφορές, και διάφορες επενδύσεις που έχουν ε, γίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Και με τα διεθνή χρηματοοικονομικά θεσμικά όργανα. Και έτσι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να μπορούν να μπουν στην υπόθεση των διευρωπαϊκών διαδρόμων και δικτύων. Ελπίζω να συνεχιστεί η καλή στενή μας συνεργασία και έτσι τα Βαλκάνια να τύχουν αυτή τη πρόσοχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας διαβεβαιώ πως η Επιτροπή μας θα είναι στο πλευρό σας στην προσπάθεια αυτή. Αλλά εάν δεν προχωρήσει η τοπική περιφερειακή οικονομική πολιτική συνεργασία τότε δεν θα υπάρξει ακριβώ ε, κάποια απορία. Αυτή είναι η λιδία λίθος. Ε, αν υπάρχει συνεργασία με τους γείτονες θα υπάρχει και συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί θα φανεί. Λοιπόν, ο κύριος Σαλαφράνκα μας ζήτησε τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς. Εκεί ήθελα να σταθώ. Σε αυτό που είπατε κι εσείς. Και ο κύριος Τσέλερ και ο κύριος Φασάκας, πρώην συναδελφός μας, τα είπανε. Ίσως μια από τις που μας επισκέπτεται. Και είπανε, λέγω, ότι έχουμε εδώ μια προοπτική θετική. Είναι δύσκολη συγκυρία. Δούμε πόσο σημαντικά είναι τα Δυτικά Βαλκάνια. Τέτοιε ώρες. Πολύ καλά τα είπατε, Πρόεδρε. Στην Ολομέλεια εγκρίναμε την έκθεση για το Μαυροβούνιο. Γιατί έχουμε στην περιοχή περίεργα συμβάντα. Έχουμε τις εκλογές και πρόκειται η Ολομέλεια να ε, αποφανθεί για τις ε, άλλες χώρες που είναι τόσο σημαντικές για την σταθερότητα της ε, Υπήρου. Όπως τα είπε ο πρόεδρος Επιτροπής, πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά τη Συμφωνίας ε, Σύνδεσης και Σταθερότητας. Ξεκάθαρα τα είπε το Ελληνικό Συνέδριο ότι περνάμε δύσκολες ώρες και χρειάζεται αυτές τις δύσκολες ώρες σημαντική οικονομική προσπάθεια. 2007-2014 ξοδέψαμε 5 δις και επομένως θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και την παρουσία μα Βάσει των αρχών μας όπω τα εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περιφερειακή συνεργασία, για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, καταπολέμηση της διαφθοράς, χρηστή διακυβέρνηση, συνεργασία. Με τίποτα να μην ε, πέσει η επιρροή μας προς αυτές τις χώρες. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη διαχείριση όλων αυτών των σημαντικών ε, ποσών που εκταμιεύουμε και αυτό να γίνει γρήγορα. Πολύ σωστά τα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας είπε τι χρειάζεται να γίνει για την προβολή του έργου μας. Έχουμε σε άλλη συζήτηση μιλήσει για το ε, πώς θα πρέπει να προβάλλεται το έργο τη κοινότητα από τα γραφεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και, και στα Δυτικά Βαλκάνια. Μια που κάνουμε τέτοια οικονομική προσπάθεια, ε, εκεί μπορούμε να βελτιωθούμε. Όπως τα λέει ο κύριος Τσέλος στο κείμενό του. Όπως τα λέει και το ελληνικό συνέδριο στη δική του έκθεση. Αξίζει τον κόπο. Καλά τα λέει η έκθεση. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Βεβαίως και έχει προβλήματα με τους ανθρώπινους πόρους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει όλοι μαζί πάντως να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε να πλαισιώσουμε αυτή τη στρατηγική προτεραιότητα και να πιάσουν τόπο όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δίνουμε στα Δυτικά Βαλκάνια. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και θα παραμείνει και για το μέλλον έτσι. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Σαβάρμα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο και κυρίως τον κύριο Φάζακας για αυτό το πολύ σημαντικό έγγραφο. Όπως και ο κύριος Σαλαφράνκο με, τόσο μεγάλη, με την εμπειρία που έχει στις εξωτερικές σχέσεις, όπως το τόνισε ο ίδιος, πρέπει να προσέξουμε την περιοχή αυτή ακόμα περισσότερο, την γεωγραφική περιοχή αυτή. Αλλά ζήτησα τον λόγο για το εξής. Μισό τη Δευτέρα το πρωί να ερχόμαστε και να λέμε τι έπρεπε να έχει γίνει πριν από χρόνια. Τους λεγόμενους προπονητές της Δευτέρας μετά τον αγώνα. Σοδεύουμε τόσα εκατομμύρια ευρώ αναχώρα 5,1 δισεκατομμύρια για το επταετές πρόγραμμα. Οπότε και εγώ ως προπονητής μετά τον αγώνα τη Δευτέρα το πρωί θα πω τα εξή. Επί 25 χρόνια κάλυψα τους πολέμους της Ιουγκοσλαβίας. Και αν ήμασταν συνεπείς και συστηματικοί στην επένδυση των χρημάτων μας στην παιδεία των μικρών παιδιών στα Βαλκάνια. Τα παιδιά αυτά που γεννήθηκαν στον πόλεμο κατά την κατάρρευση της χώρας τα παιδιά αυτά αναλαμβάνουν τώρα την ευθύνη τους στις κοινωνίες τους και σε λίγα χρόνια θα βρίσκονται σε αποφασιστικές θέσεις στις εκάστοτε χώρες τους Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Με τους λίγους πόρους που μπορούμε να επενδύσουμε σε κάθε μία από τις χώρες αυτές θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη διαφορά στοχεύοντας καλύτερα επειδή εάν απλά διασπείρουμε τα χρήματα, τα πετάξουμε στον αέρα τότε κάποια κέρματα θα πέσουν στον καθένα, το υπόλοιπο θα το πάρει η γραφειοκρατία, αλλά έτσι δεν θα επιτύχουμε τίποτα. Μετά από άλλα 25 χρόνια θα είμαστε εδώ και θα λέμε τα ίδια. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ποτέ δεν είναι αργά για να αρχίσουμε. Και πιστεύω πως πρέπει να συγκεντρωθούμε στη δημιουργία μιας βάσης. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε έναν ασθενή που, έχει, που μεγαλώνει ήδη με καρκίνο εδώ και δεκαετίες. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον και να μεγαλώσουμε την επόμενη γενιά σε αυτή την περιοχή του κόσμου και πρέπει να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης μας, αν μας ενδιαφέρει το δικό μας μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Για αυτό που είπες με τους προπονητές μετά τον αγώνα. Αυτή η Επιτροπή ήταν ο τελευταίος οπαδός της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανασυγκρότησης. Νομίζω υπόκειτο στην Επιτροπή επειδή υλοποίησε πολύ γρήγορα έργα μετά τον πόλεμο μετακαταργήθηκε υπό συνθήκες αδιαφάνειας αλλά Εάν έβλεπε κανείς τα προβλήματα και θυμάμαι τις αρχές της θητείας μου εδώ στην Επιτροπή αυτή όταν ακούγαμε τις εκθέσεις του οργανισμού αυτού τι προβλήματα υπήρχαν τότε. Δεν υπήρχε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Φρόντιζε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση για την τροφοδοσία του Κωσυφοπαίδου με ηλεκτρικό ρεύμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα τεράστιο σκάνδαλο. κτίζαμε διαμερίσματα για ανθρώπους. Οι συνθήκε ήταν τόσο άσχημε για τους ανθρώπους στα Βαλκάνια, στις επιμέρους χώρες διαφορετικές βέβαια. Είχαμε τα προβλήματα μεταξύ των διάφορων εθνοτικών ομάδων και σήμερα σε σχέση με τότε οι συνθήκες είναι σχεδόν παραδεισιακές Φυσικά και εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι με ένα τέτοιο παράδεισο επειδή έχουμε περαιτέρω σχέδια. Θα ήθελα να ταχθώ υπέρ του να δούμε και τι επιτύχαμε. Και επιτύχαμε πολλά. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα στα Βαλκάνια οι συνθήκες θα ήταν ακόμη πιο καταστραφικές. Συζητούμε λοιπόν προβλήματα σε πολύ ψηλότερο επίπεδο από ό,τι τότε. Και αυτό είναι αλήθεια. Θα ήθελα να το αναφέρω ώστε να μην πάρει η συζήτηση εσφαλμένη κατεύθυνση. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι περήφανη για αυτό που κατάφερε, αλλά δεν πρέπει να επαναπαθεί, επειδή απομένει πολλή δρόμο. Πιστεύω πως το ζήτημα της συμφιλίωσης των εθνικών ομάδων θα συνεχίσει να είναι ένα σημαντικό ζήτημα και όπου θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες ακόμα και για μικρή πρόοδο. Έχουμε, ακούμε διαφορετικά πράγματα από εκεί αλλά έχουμε ένα σαφές καθήκον. Γι' αυτό και θα ήθελα από σήμερα να ταχθώ υπέρ του η παρούσα επιτροπή να στείλει τουλάχιστον μια επταμελή αποστολή το καλοκαίρι εκεί. Επειδή αν το κάνουμε όπως στην Πολωνία τον Απρίλιο, εκεί είμαστε τρεις. Λοιπόν, θα ήθελα αγαπητοί συναδελφοί να σας ζητήσω ελάτε μαζί στην Πολωνία. Πώς μπορούμε να, να επισκεφτούμε τον το κράτος που παραλαμβάνει τις περισσότερες διαφορετικές βοήθειες με μια τόσο μικρή αποστολή. Εάν είναι έτσι καλύτερα να σταματήσουμε. Παρακαλώ, θα στείλω και ένα email αργότερα. Περιμένω πως τα μέλη εδώ πέρα θα δείξουν κάποιο ενδιαφέρον για, τον, για το κράτος που παραλαμβάνει τις μεγαλύτερες βοήθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και αν είναι η εβδομάδα μετά το Πάσχα, όταν πολλοί από εμά θα προτιμούσαν ίσως κάποιο πιο ζεστό κράτος, κάποια χώρα πιο κατάλληλη για διακοπές. Παρακαλώ πολύ αποφασίστε το επειδή είμαστε μόνο τρεις άνθρωποι αυτή τη στιγμή επειδή τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας και οι άνθρωποι βασίζονται σε εμά. Πάντα συνεχίζουμε, παίρνουμε αλληλογραφία, πολλή αλληλογραφία από οπαδούς μας. Παίζουμε έναν ρόλο σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Μια διαφήμιση ήταν αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Μότον, θέλετε να πάρετε το λόγο ή αποχωρείτε ευχαριστημένος που επιζήσατε. Είστε ικανοποιημένο λοιπόν. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον συνάδελφο Φάσακα. Ο συνάδελφο Τσέλερ θα πάρει το λόγο όσον αφορά τη διαφήμιση της Πρόεδρου. Ίσως πρέπει να σκεφτούμε πως όταν πηγαίνουμε σε χώρες όπως την Πολωνία που βρίσκονται πολύ κοντά εάν δεν μπορούμε ίσως κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων να στείλουμε μια αποστολή και όχι μόνο σε μια πράσινη εβδομάδα, επειδή τότε μας ρωτάνε όλες οι επιτροπές αν θέλουμε να πάμε κάπου. Όσον αφορά το θέμα των δυτικών Βαλκανίων, ο κύριος Αλαφράνκα είπε ήδη κάποια πράγματα τα οποία είναι απολύτως σωστά. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αλλά όταν κοιτάω τις πολιτικές συνθήκες και τους πολιτικούς παράγοντες εκεί, τότε εξασθενεί λίγο η ελπίδα μου. Ίσως θα πρέπει να θυμόμαστε αυτό που είπε και ο Πέτρης Αδάρμα, πως πρέπει να βρούμε να επιλέξουμε καλύτερα νέους τομείς δραστηριοποίησης, να ενισχύσουμε τα προγράμματα Εράσμους για τους νέους στα Βαλκανικά αυτά κράτη και ίσως να αρχίσουμε μια επικοινωνιακή στρατηγική για να είμαστε παρόντες στα επιτόπου μέσα μαζικής ενημέρωσης για να δείξουμε επιτόπου τι έχει γίνει μέχρι στιγμή, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή έτσι ώστε οι άνθρωποι επιτόπου να μην χάσουν την πίστη σε εμάς επειδή εκεί αυτή τη στιγμή όλα είναι πολύ δύσκολα αν βασιστεί κανείς αποκλειστικά στους πολιτικούς παράγοντες. Αυτό το να διατηρηθεί η πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πολύ σοφή ρίση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Πιστεύω ότι μια έκθεση είναι έτοιμη που περιμένει την παρουσίασή της. Είναι αυτή του Μόλδαβα εκτός μικροφωνού είναι η προσέγγιση hotspot εργάζομαι επί μιας εργασίας για την Τουρκία την τελευταία εβδομάδα είχα τη δυνατότητα να μείνω στην Άγκυρα όπου και υποδέχθηκα από όλα τα μέλη της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου που ενδιαφέρονται ακόμα σε μια, για μια στενή συνεργασία και για το μέλλον της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και εξεπλάγει ιδιαίτερα πως τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι από, σε μια εκδήλωση της Επιτροπής των Περιφερειών είδαμε πως όλες οι χώρες που εκτιμούν το έργο αλλά θεωρούν πως οι πόροι δεν είναι αρκετοί. Γι' αυτό πάντα λένε ότι θα μπορούσαν να έχουν πάρει περισσότερα. Έχετε δίκιο λοιπόν. Πρέπει να τους επιστήσουμε την προσοχή πως δεν είναι δωρεάν λεφτά αλλά είναι χρήματα τα οποία δίνονται για να σας βοηθήσουν να φέρετε τις χώρες σας στο ύψος των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως είπατε, ο πολιτικός διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί, έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να επενδύονται αποτελεσματικά στην βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαρίστω τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο θα ξαναπάω στο Βελιγράδι. Ευχαρίστω και από πλευρά μα, οπότε ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό τη υπηρεσία διάταξη. Θεωρώ δεδομένο πω θα σα ξαναδούμε, οπότε δεν σα αποχαιρετώ. Θα ήθελα ωστόσο να σα ευχαριστήσω για την έκθεση και τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ επίση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελειώνουμε το σημείο 6, περνούμε στο σημείο 7 μελέτη με θέμα συγκρούσει συμφερόντων σε κρατημέλη σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης κατά τη διαχείριση χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λόμαϊερ, Χένεκε, Πίκη και Μόιλανεν είναι οι συντάκτες. Die Frau Kollegin η συγκήτρια είναι η κυρία Λαμπάγιοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκπρόσωπη της Bloma Sands, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το θέμα μας αφορά τους κώδικες συμπεριφοράς και τη συγκρούση συμφερόντων σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης ε, των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων, κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Η ανάγκη διαφάνειας ε, της ε, δημοσίας διοίκησης στο εθνικό και ενωσιακό επίπεδο είναι βασική ε, αναγκαιότητα για να μην υπησέρχονται προσωπικά συμφέροντα στην διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Νομίζω λοιπόν πως η ανάγκη διαφάνειας έχει γίνει αντιληπτή τα τελευταία χρόνια όταν επιτυχημένοι επιχειρηματίες ε, κατεβαίνουν ε, στην πολιτική όπως και εγώ άλλωστε από τις επιχειρήσεις ήρθαν στην πολιτική και είναι ενδιαφέρον το να βλέπω το που πηγαίνουμε σε αυτά τα ζητήματα γρήγορα λοιπόν το θέμα αυτό έχει μελετηθεί και αναλυθεί ήδη πολλές φορές ε, το 2005 ο ως δημοσίευσε μια εργαλειοθήκη που λέγεται Διαχείριση Συγκρούσεων Συμφερόντων στο Δημόσιο Τομέα. Το 2007 η Κομισιόν έκανε μια συγκριτική μελέτη που αφορά ακριβώς τους τρόπους διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων για αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2008 η μονάδα αξιολόγησης του ΔΕΛΤΑΝΗ ΤΑΦ δημοσίευσε μια σχετική μελέτη. Το 2009 η Επιτροπή μας ε, μελέτησε ακριβώς τον κώδικα συμπεριφορά των επιτρόπων για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και το 2012 το Πανεπιστημίο της Βασιλείας μελέτησε το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων στην παγκόσμια δημόσια και εταιρική διοίκηση. Υπάρχουν πολλά πράγματα λοιπόν. Ζητήσαμε ως Επιτροπή αυτήν την μελέτη γιατί θέλουμε να αναλύσουμε και να συγκρίνουμε τους υφιστάμενους κώδικες συμπεριφοράς που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο της κοινή διαχείρισης των οικονομικών της Ένωσης. Η μελέτη επίσης ε, μας λέει κάποια πράγματα για την πιθανή ύπαρξη νομοθεσίας ε, της ρύθμισης ε, του ζητήματος και του εάν οι κώδικες συμπεριφοράς είναι ο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Και επίσης ζητήσαμε να βρεθούν οι βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο που προκύπτουν από τις αναλύσεις της κατάστασης. Αυτός ήταν ο στόχος. Θεωρώ πως η μελέτη ανταποκρίθηκε στους στόχους και ευχαριστώ να δώσω τον λόγο στους συντάκτες. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις γιατί θα ήθελα να πάω εις βάθος σε κάποιες δήματα, οπότε θα αφήσω τις ερωτήσεις μου για μετά την παρουσίαση αν μου επιτρέπετε ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ οπότε τον λόγο έχουν οι συντάκτες της μελέτης ποιος θα ξεκινήσει ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την μελέτη με τίτλο «Κώδικες συμπεριφοράς και συγκρούσεις συμφερόντων» σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης ε, της διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων. Στόχος είναι να καταλάβουμε πώς οι διοικήσεις των ε, κρατών μελών που εμπλέκονται στην διαχείριση των κονδυλίων αυτών διασφαλίζουν την διαφάνεια. Σήμερα λοιπόν η παρουσίασή μας έχει τέσσερα τμήματα. Θα κάνουμε μια παρουσίαση του περιεχομένου και μετά οι συνάδελφοι θα παρουσιάσουν τα ευρήματα, τις βαλίτσες πρακτικές και τις συστάσεις. Και βεβαίω αναμένουμε και τις ερωτήσεις σας. Μάλιστα, ωραία. Η μελέτη διεξήχθη μεταξύ 2000 και 2017 περιείχε σημαντικά στοιχεία, καλύψαμε και τον νόμο και το soft law, τα θέματα της ακεραιότητας, εξετάσαμε τα ζητήματα εκείνα της ακεραιότητας και τα επίπεδα εκείνα τα οποία πιθανότερα είχαν κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Το πλαίσιο αυτό λοιπόν αφορούσε την κοινή διαχείριση κοινωτικών κονδυλίων και συγκεκριμένα το ΕΤΠΑ και το Κοινωνικό Ταμείο. Εστιάσαμε στην σύγκριση συμφέροντων που αφορά τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Και ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο, οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από εκπροσώπους ενδιαφερομένων και των ταμείων των διαρθρωτικών και των επενδυτικών ταμών και είναι από τις εθνικές ε, περιφερειακές αρχές αλλά και θεματική ειδική στα επιχειρησιακά προγράμματα έρευνα, κοινοτομία, φύλλο, περιβάλλον και βεβαίως ε, το θέμα. Αυτό ευθυγραμμίζεται πολύ συγκεκριμένα με το ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο ε, πρέπει να εμποδίζει την σύγκρουση αυτή των συμφερόντων. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ένα μέλος μια επιτροπή παρακολούθησης που εκπροσωπεί π.χ. μια περιφερειακή ένωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως κοινωνικός εταίρος και ταυτόχρονα έχοντας μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να έχει μια σύγκριση συμφερόντων εάν σχεδιάσει την προκήρυξη έτσι ώστε να ευνοεί την δική του επιχείρηση. Οπότε ακριβώς αυτή είναι η σύγκρουση συμφερόντων που ενδιαφέρει τους ε, συμμετέχοντες και μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει ιδιαίτερη ε, προσοχή. Εστιάσαμε λοιπόν σε τρία βασικά ερωτήματα, δηλαδή το τι υπάρχει από πλευράς ε, πολιτικής σύγκρουση συμφερόντων στην κοινωτική χρηματοδότηση και στην κοινή χρηματοδότηση για αν λειτουργεί και τι πρέπει να γίνει. Κάναμε λοιπόν συνεντεύξεις με ναι, ενδιαφερομένους ε, έρευνα των εθνικών αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση κοινωτική χρηματοδότηση και βεβαίω και κάποια περιπτωσιολογία. Είχαμε λοιπόν την Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο, απασχόληση, τον Όλαφ, τον Διαμεσολαβητή και οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών. Στοχεύσαμε επίσης συγκεκριμένε διαχειριστικέ αρχέ. λάβαμε απαντήσει από 17 κρατημέλη, βλέπετε τις ε, Χώρε ε, που έλαβαν μέρος ε, και απάντησαν στη δεύτερη ερώτηση εάν λειτουργεί. Εστιάσαμε σε 7 κράτη-μέλη, κάναμε συνεντεύξεις και έρευνα γραφείου και βεβαίω ε, αυτά σε συνεργασία με τον ΕΟΧ και της Φορικής Ναυηγίας. Η έννοια λοιπόν αυτή περιλαμβάνει την ρυθμιστική βάση όπως αυτή αναφέρεται στις κατευθυντήρες γραμμές. Η Κομισιόν λοιπόν έχει εκδώσει κάποια έγγραφα στρατηγικής ε, και κατευθυντηρίων γραμμών και αξίζει να σημειώσουμε πως ε, η άκρηση τη εμφάνιση των συγκρούσεων συμφερόντων βλέπουμε εδώ πέρα, παραδείγματο χάρη, ότι η κοινή στρατηγική καταπολέμηση απάτη 2010-2011 δεν αναφέρει την έννοια αυτή, ενώ οι επόμενες στρατηγικές να αναφέρουν όπως και τα περισσότερα έγγραφα κατεύθυνση. Επίσης, τα έγγραφα αυτά κυρίως αναφέρονται στο ζήτημα στο πλαίσιο των δημοσίων προμηθειών. Οπότε υπάρχουν λίγες και έμεσες αναφορές σε τέτοιες καταστάσεις εκτός των ε, δημοσίων προμηθειών. Και πράγματι οι πληροφόρες που λάβαμε, η ανάδραση ήταν πως ε, υπάρχει μια συνοχή στο θέμα της πρόληψης απάτης και της, των δημοσίων προμηθειών. Αξίζει λοιπόν να σημειώσουμε πως υπάρχουν κάποιες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πληροφόρηση που ε, ενημέρωσαν 1.500 ενδιαφερόμενους σε σεμινάρια στις χώρες και βλέπουμε ότι οι αντιδράσεις ε, των κρατών μελών ε, αφορούσαν κάποιες ε, κατευθυντήριες ε, γραμμές. Θα τα πει ο Κριστόφ. Χαίρομαι που τα συζητούμε τώρα. Να σας πω τι γίνεται με αυτή την έρευνα. Πρώτα να σας πω δύο λόγια όσον αφορά την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των πολιτικών για τις σύγκριση των συμφερόντων και επιτρέψτε μου να σας πω πρώτα τα εξής. Ο υποφαινόμενος εδώ και μια δεκαπενταετία ασχολείται με το θέμα. Και τότε ασχοληθήκαμε με το θέμα και τότε ήταν κάτι το αφηρημένο, κάτι το φιλοσοφικό. Δεν, δεν υπήρχε ε, σχετική νομοθεσία. Επιτροπές ε, ελέγχων, επιτροπές ε, ηθικής, νομοθεσία και τότε το ηθικό αυτό θέμα, η ηθική ακεραιότητα, αλλά κυρίως, κυρίως η σύγκρουση πρώτων ε, ξεκίνησε. Ήταν μια έκρηξη μπορούμε να πούμε και τώρα βλέπουμε να υπάρχουν ε, νόμοι διεθνώς και σε επίπεδο ένωσης και σε εθνικό επίπεδο και τα έχουμε δει αυτά και σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό επομένως δεν μας λείπουν τα νομοθετήματα. Και έχουμε και τους κώδικες διοντολογίας ε, που δεν έχουμε τώρα τον χρόνο να το συζητήσουμε και ήταν τα τελευταία χρόνια ότι όλο ένα και πιο δημοφιλή γίνανε όλα αυτά. Δεν υπάρχει τώρα κανένας οργανισμός, ε, κυβέρνηση, επάγγελμα που να συνεχίζει την ύπαρξή του χωρίς κάποιο κώδικα διοντολογίας. Επομένως μιλούμε για έκρηξη του τομέα αυτού. Πολλές φορές βέβαια, αυτά είναι νεκρό γράμμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η αποτελεσματικότητα αυτών των κώδικων διοντολογίας. Αν πιάνουν τόπο δηλαδή όσον αφορά τη σύγκρουση συμφέροντων και την καταπολέμηση. Οπότε έχουμε διάφορε εργαλειοθήκε, κατευθυντήριες γραμμές και μιλούμε για πάρα πολλές τέτοιε εργαλειοθήκες που υπάρχουν που πριν 15 χρόνια δεν υπήρχαν. Όπως η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Υπέροχο. Γραφτό αλλά το ίδιο ισχύει και για τις επιτροπές ελέγχου για των σχετικών υπαλλήλων που υπάρχουν παντού. Σχετικά, νέα εξέλιξη είναι αυτό. Τώρα, κεντρώνουν την προσοχή του στα θέματα εφαρμογής. Παλιά ήταν μια συμβολική πολιτική. Ε, εγκρινόταν ένας ε, κώδικας, ένας κανονισμός, ένας νόμος και εκεί σταμάταγε η υπόθεση. Τώρα όμως διαπιστώνουμε άλλη τάση. Εστίαση στην εφαρμογή. Πράγμα σοβαρό αυτό για το τι θα πρέπει να διέπει η διαφάνεια. Περισσότερη διαφάνεια επομένως έχουμε από στο παρελθόν. Κάλυψε από τα ΜΜΕ. Να το δίλημα. Περισσότερα ΜΜΕ, περισσότερα περισσότερη διαφάνεια, από την άλλη μεριά όμω περισσότερη σκανδαλολογία. Οπότε είναι το θέμα πια τη εμπιστοσύνη ή τη δυσπιστία. Και ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα, στο θέμα τη αποτελεσματικότητα. Γιατί είδαμε την τελευταία 15 ετία ότι οι πολιτικέ <coughs> και η νομοθεσία για την σύγκρουση συμφερόντων έχουν πάρει περισσότερη σημασία και είναι πιο δημοφιλή σε πολλές χώρες δεν υπάρχει τρομερά έντονη δραστηριότητα γι' αυτό και τελείως διαφορετικό βέβαια είναι το θέμα του πώς οι πολιτικές μας θα είναι αποτελεσματικές πώς θα μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτό είναι άλλη ιστορία αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιεύσεις αλλά και μελέτες δεν έχουμε στοιχεία για το ότι έχει συγκρατηθεί η διαφθορά μάλλον αυξάνεται άρα Πάμε τώρα στο πώς θα γίνουν πιο αποτελεσματικά τα σχετικά πλαίσια. Νόμοι, κώδικες, όσο περισσότερα θέματα θεωρούνται ως σύγκρουση συμφερόντων, ε, τόσο περισσότερη νομοθεσία θα υπάρχει, αλλά και πολιτικές. Και νομίζω συμφωνούμε ότι αυτό από μόνο του είναι θετικό. Αλλά βέβαια έτσι αυξάνεται και η παραβίαση των σχετικών κανόνων. Άρα θα έχουμε περισσότερες σχετικές εκθέσεις, αναφορές, δημοσιοποίηση, ε, δημοσίευματα για σκάνδαλα, δυσπιστία. Άρα το θέμα είναι το πώς θα αναβαθμίσουμε την αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Όμως η πολιτική για την ε, σύγκρουση συμφερόντων βέβαια είναι μια πολιτική της δυσπιστίας. Για να πάμε επομένω να προστατεύσουμε την ε, ακεραιότητα. αλλά να δούμε το πώς δεν ε, θα φουσκώσουμε αυτή τη δυσπιστία γιατί έχουμε όλο ένα περισσότερες ε, παραβάσεις των υπαρχουσών διατάξεων. Επίσης αυτοί οι κώδικες διοντολογία είναι πολύ δημοφιλείς για τους πολιτικούς, τους υπαλλήλους, δημοσίου υπαλλήλου, για κάθε επάγγελμα, για κάθε κλάδο. Όμως ακόμα εκκρεμούν πολλά ερωτήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του. Για να δούμε τώρα τι άλλο λέει η μελέτη και η έρευνά μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων ποιο είναι η γνώση της διάστασης του προβλήματος. Δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να σας πούμε. Το έχουμε ψάξει πολύ, αλλά τελικά πολύ λίγες ενδείξεις και αποδείξεις βρήκαμε και στοιχεία. Γιατί μέχρι σήμερα υπάρχει πολύ περιορισμένος έλεγχος και εποπτεία σε αυτό. Έχουμε νομοθεσία που συνεχώς ε, επεκτείνεται όσον αφορά την ε, διαφθορά. Είναι πικάντικο και σεξι και δημοφιλές, αλλά για τη σύγκρουση συμφέροντων δεν έχουμε τόσο μεγάλη δραστηριότητα. Όχι, είπε η Όλαφ όταν ρωτήσαμε. Δεν παρακολουθούμε τη σύγκρουση συμφέροντων. Το ίδιο είπαν και τα κράτη-μέλη. Οι περιφερειακές αρχές, τοπικές αρχές. Όλοι αρνητικά. Ε, αυτό είναι το θέμα τώρα με τους πόρους στις επιτροπές εποπτείας. Αυτό είναι ακόμα αρμοδιότητα της ε, κάθε επιτροπής. Πρόκειται για αυτορύθμιση. Όμως δεν πιάνει τόπο αυτό, δεν αποδίδει. Ας πούμε έχουμε συνεντεύξεις, έχουμε επιτόπου δουλειά, έξω και όχι θεωρητικά με στοιχεία. Ήρθαμε σε επαφή με πρόεδρο των Επιτροπών, αυτή ήταν πολύ γενικοί, μας είπαν τους κανόνες διαδικασίας, της λειτουργίας και όλοι αυτοί οι κανόνες, περισσότερες περιπτώσεις δηλαδή, μιλούσαν για σύγκρουση συμφερόντων. Όμως, άλλο τελείωσαν το θέμα όταν έρχεται η ώρα να συζητηθούν, να εφαρμοστούν ε, για να επιβληθούν οι σχετικοί κανόνες και επομένως ε, τα στοιχεία δείχνουν ότι σε περισσότερες επιτροπές και χώρες ότι εξετάσαμε δεν υπάρχει εφαρμογή, υλοποίηση παρά τους τόσο στεγανούς τέλειους ε, κανόνες. Άρα, στην καθημερινή λειτουργία των Επιτροπών αυτά δεν συζητιούνται. Πολύ λίγα είναι τα πρωτόκολλα που δημοσιοποιούνται για το ότι σε μια μέρη σε διάταξη θα ζητηθεί στην Επιτροπή η σύγκρουση συμφερόντων και το τι θα γίνει αν έχουμε σύγκρουση συμφερόντων, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει. Επομένως η μελέτη μας κατέληξε στο ότι η αυτορύθμιση δεν ισχύει. Θα πρέπει να υπάρχει ε, εποπτεία από ανεξάρτητους φορείς. Θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Πρωτόκολλα, διαφάνεια για τις αποφάσεις των επιτροπών και με, που αυτά ακούγονται πάρα πολύ ακαδημαϊκά αλλά θα πρέπει να Υπάρχει περισσότερη συνειδητοποίηση του προβλήματο. Θα πρέπει αυτό να τον αναλάβει ο κάθε πρόεδρο, κάθε επιτροπή, Εφαρμογή των διαδικασιών. Και αυτά πρέπει να αντιμετωπίσει. Πολύ συχνά όμω δεν τα κουβεντιάζουν αυτά οι πρόεδροι και οι επιτροπές. Τα τη σύγκρουση συμφερόντων. Οπότε και αναδύεται το ερώτημα γιατί δεν συζητιούνται οι σύγκρουσει των συμφερόντων. Ε, πολλέ φορέ όχι γιατί είναι κακοί άνθρωποι θέλουν να αποφύγουν το στρίμωγμα, αλλά πολλές φορές οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών υποτιμούν το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόβλημα. Οπότε βρίσκουν το θέμα περίπλοκο, ακαθόδες, το ανέχονται. Άλλωστε τρώει και χρόνο, γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες για να συζητήσουν. Ε, συνέπεια είναι ότι δεν συζητιούνται συγκρούσεις συμφέροντων. Έχουν ευθύνες οι πρόεδροι. Οι πρόεδροι θα πρέπει να τις αναλάβουν αυτές τις ευθύνες τους. Υπάρχει περισσότερη συνειδητοποίηση του προβλήματος. Έτσι ολοκληρώνουμε επομένως... τον προβληματισμό μας ότι στον πολιτικό βίο Όσον αφορά την νομική δραστηριότητα, το θέμα μας έχει υποστεί πολύ μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί τώρα έναν τομέα πολιτικής, όπου πάρα πολύ εντατική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί. Όταν όμως έρχεται η ώρα των επιτροπών, των διερωτικών ταμείων, η πραγματικότητα είναι όλος διαφορετική. Δεν συζητιέται το θέμα. Ευχαριστώ. Um, yeah, uh, thanks also from my side for having us here. Uh, and I'm... Ευχαριστώ επίσης από πλευράς μου που μας υποδεχθήκατε εδώ. Θα συνεχίσω την ανάλυση του Κρίστοφ Λέμκε και θα υπογραμμίσω κάποιες από τις καλές πρακτικές που συγκεντρώσαμε για τη μελέτη μας. Πιστεύω πως πρέπει λίγο να προχωρήσουμε στις διαφάνειες Τώρα μιλούμε για την διαφάνεια 9, εάν ο υπεύθυνο θα μπορούσε να προχωρήσει. Ο τίτλος είναι «Καλές πρακτικές». Πάμε λοιπόν. Όπως ακούσαμε, υπάρχει λίγη γνώση, λίγη ευαισθητοποίηση, ιδίως σε περιπτώσεις που έμοιαζαν θετικά παραδείγματα βρήκαμε ενταξιακές προσεγγίσεις δηλαδή τη συμπερίληψη εξωτερικών ειδημόνων και αξιολογήσεων για τους κινδύνους και τα επίπεδα έκθεσης των προγραμμάτων και για την άμεση αντιμετώπιση των εντοπισμένων αδυναμιών στο σύστημα ελέγχου. Με το στόχο αυτό είναι σημαντικό να ενισχυθεί επίσης ο μηχανισμός πρόληψης των κινδύνων και έτσι να προληφθεί η κακή πρακτική με μέσα όπως μια πολιτική πληροφοριοδοτών που σε πρώιμο στάδιο θα μπορούσε να εντοπίσει απειλές και κινδύνους. Τρίτον, Ήδη τονίστηκε πως είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο η καταγραφή των ιχνών όλων των αποκλήσεων από τις τυπικές διαδικασίες που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες όλων τον κύκλο του προγράμματος. σε ένα τέτοιο σύστημα περιλαμβάνεται οποιαδήποτε απόκληση, είτε αυτή οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων είτε όχι. Επειδή αυτό θα προκαλούσε επίσης μία από τις δυσκολίες, δηλαδή την έλλειψη γενικής παρακολούθησης. Θα μπορούσε να μας δώσει ένα εργαλείο για μία επισκόπηση δυνητικών περιπτώσεων, πώς αντιμετωπίζονται. Θα ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο να υπάρχει. Επίσης διαπιστώσαμε μια ανάγκη εσωτερικών διαδικασιών αναθεώρησης όσον αφορά παρατυπίες, σε συνδυασμό επίσης με ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο και αξιολόγηση προγραμμάτων. Δηλαδή συνδεδεμένοι ανεξάρτητοι δήμονες ήταν ένα σημαντικό βήμα. Επίσης πρέπει να γίνεται καλύτερη παρακολούθηση των προγραμμάτων επιτόπου ιδίως σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, όπως προκαθορισμένα προγράμματα, με διαφορετικές διαδικασίες όσον αφορά την επιβράβευση. Επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τους ανθρώπους που εργάζονται επί των έργων στην άλλη άκρη, στην άκρη του αποτελέσματος. Με τέτοια προσέγγιση θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα κατά την εφαρμογή προγραμμάτων και να αναπτύξουμε από τη γνώση των προβλημάτων καινοτόμα, καινοτόμους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε μελλοντικές συγκρούσεις συμφερόντων. Από τις καλές πρακτικές αυτές περνούμε σε κάποιες συστάσεις. Θα είναι η επόμενη διαφάνεια. Βρήκαμε πως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του EA χρήσιμο εργαλείο ήταν ο διορισμός ενός διαχειριστή κινδύνων αρμόδιου για προβλήματα για τομείς ή για επιμέρους προγράμματα ο οποίος θα παρακολουθεί όλο τον κύκλο του προγράμματος από την επιλογή ως την αξιολόγηση για να έχει τη συνολική γλώσση. Φυσικά η δημόσια αποκάλυψη σημαντικών επιχειρηματικών ή χρηματοπιστωτικών οικονομικών συμφερόντων σε μια δημόσια βάση δεδομένων ή ένα δημόσια προσβάσιμο μητρό. Επίσης, εσωτερικές και εξωτερικές παρουσιάσεις για την ευαισθητοποίηση για, τους για τον αντίκτυπο των συγκρούσεων συμφερόντων. Επίσης, ευαισθητοποίηση για την φύση και την... τον δυνητικό αντίκτυπο περιπτώσεων σύγκρουση συμφερόντων. Μπορεί να μοιάζει αμεληταίο, αλλά στο τέλος ε, δημιουργείται μια συγκεκριμένη δυναμική που αυξάνει τον αντίκτυπο. Ενημέρωση σε όλα τα πρωτόκολλα, σε όλες τις διαδικασίες. Αναφέρομαι σε πρωτόκολλα τα οποία θα πρέπει να αναθεωρούνται, να εξετάζονται ανεξάρτητα. Περνούμε μετά σε μια εστίαση στην ακαιρεότητα. Η ηθική ηγεσία είναι η κλειδί εδώ. Θέλουμε να, να τους ανθρώπους να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να συμπεριφερθούν με τρόπο ώστε να συμμορφώνεται σε μια κουλτούρα επιχειρηματική και οικονομική. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την κουλτούρα αυτή και να συμπεριλάβουμε εξωτερικούς ειδήμονες και θα πρέπει να γίνεται τακτική εκπαίδευση και ενημέρωση επειδή όπως προχωρά η κοινωνία μας όχι μόνο σε τεχνολογικό επίπεδο προκύπτουν όλο ένα και νέοι, νέες συγκρούσεις συμφερόντων δεν μπορούμε να έχουμε ένα σταθερό σύνολο κανόνων το οποίο δεν προσαρμόζεται στις νέες προκλήσεις Πιστεύω πως αυτές είναι οι κύριες συστάσεις που θα ήθελα να δώσω εδώ. Φυσικά στην έκθεση έχουμε κάποιες περισσότερες και ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τις πολύ ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις. Είναι περισσότερα από ό,τι περίμενα. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πιστεύω πως θα πρέπει να, να καταρτήσουμε έναν οδηγό βέλτιστων πρακτικών. Το λόγο έχει η εισηγήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που εκτιμάτε την μελέτη επειδή ήταν πολλή εργασία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Κάνατε πολύ καλή δουλειά και πιστεύω πως, πρέπει, πως εισέρχεται εις βάθος σε κάποια ζητήματα. Έχω συγκεκριμένες και εις βάθος ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τις απαντήσεις σήμερα, αλλά πρόκειται για ζητήματα τα οποία είδα στη μελέτη όταν τη διάβαζα πολύ προσεκτικά. Πρώτον λοιπόν, στη σελίδα 53, σημασία δεν έχει η σελίδα, δείχνεται πως μπορεί να υπάρχει μια συσχέτιση του επίπεδου σύγκρουση συμφερόνων και της εμπιστοσύνη σε δημόσιου θεσμούς. Ενώ στις σκανδιναβικέ χώρες έχουμε υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνη, γι' αυτό μπορούν να χρησιμοποιήσουν σχετικά ήπιους μηχανισμούς, όπως εθελοντικές συμφωνίες, κώδικες ή κατευθυντήριες γραμμές. Κατά την άποψή σας, ποια βήματα πρέπει να γίνουν για να αλλάξουν τα κατά μέσον όρο υψηλά επίπεδα έλλειψης εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ εύκολη ερώτηση. Ε, θα... θα... Τέσσερις ερωτήσεις θα κάνω. Περιμένετε. Η δεύτερη, λοιπόν. Στη σελίδα 54 της μελέτης ε, αναφέρεται κάποια πράγματα που είπε η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και ένα συμπέρασμα που λέει λόγω των μειωμένων αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της διαφοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει περιορισμένα μέσα όσον αφορά τα ταμεία αυτά. Τι προτείνεται για να αυξηθούν οι αρμοδιότητες της Ένωσης χωρίς να θεωρηθεί παρέμβαση στην εθνική κυριαρχία γιατί υπάρχει όπως ε, ξέρετε αυτή η ισορροπία που πρέπει να σεβόμαστε οπότε η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν πρέπει να θεωρείται παρέμβαση στην ε, κυριαρχία των κρατών μελών η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας είναι αρμοδιότητα της κοινότητας πρέπει να βρούμε την χρησιτομητή άποψη έχετε η τρίτη μου ερώτηση θα ήθελα εδώ πέρα να αναφέρω το συμπέρασμα που βγάζετε στη σελίδα 65 Επιπλέον, λέτε, μπορεί οι κώδικες να χρησιμεύουν μόνο στα άτομα εκείνα τα οποία θέλουν καθοδήγηση γιατί θέλουν να συμπεριφερθούν ηθικά. Ωραίο αυτό, αλλά δεν είναι χρήσιμο. Εάν ο αξιωματούχος θέλει να δράσει ανήθικα, είναι μάλλον απίθανο να τον εμποδίσει ένας κώδικας συμπεριφοράς. Θεωρείτε ότι το μέλλον της καταπολέμησης των συγκρούσεων συμφερόντων είναι κώδικες ε, αντί για όλο και περισσότερη και περίπλοκη νομοθεσία. Και τελευταία ερώτηση, μια δύσκολη ερώτηση, συγκεκριμένη. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Ποια είναι η άποψή σας για έναν νέο ορισμό της σύγκρουση συμφερόντων στο άρθρο 57 του ε, νέου δημοσιονομικού κανονισμού που αναφέρεται ανοίγουν εισαγωγικά για τους σκοπούς της παραγράφου 1, σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν η αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων ενός ε, ατόμου ή ε, χρηματοοικονομικού φορέα πλήττεται για λόγους ε, οικογενειακούς, συναισθηματικούς, πολιτικής ή εθνικής ταυτότητας ε, και οποιοδήποτε άλλου κοινού συμφέροντος ε, με τον δικαιοχό. Δεν υπάρχει ορισμός ε, της οικογένειας, δεν υπάρχει ορισμός του τι εννοούμε ιδεολογική συγγένεια ή εθνική συγγένεια. Ο όρος οικογένεια καλύπτει και μακρινούς συγγενείς και δεν τους έχουμε δει ποτέ. Η ιδεολογική συγγένεια καλύπτει και τις πολιτικές απόψεις κάποιου χωρίς να είναι μέλος κόμματος και όταν μιλάμε για ε, εθνικούς δεσμούς ε, σημαίνει ότι οι υπάλληλοι της Κομισιόν της χη δεν θα πρέπει να μπλέκονται σε υποθέσεις του κράτους αυτού. Ποια είναι η άποψή σας ε, για τον ορισμό της σύγκρουσης συμφερόντων. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολες οι ερωτήσεις, αλλά ως συγγήτρια έχω διαβάσει πολλές φορές την ε, μελέτη αυτή και αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα που είδα και θα ήθελα να μπω λίγο σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Είναι περίπλοκες ε, και σημαντικές ερωτήσεις. Θα απαντήσω εγώ στο πρώτο, στο τρίτο και το τέταρτο τόμο. Θα απαντήσει δεύτερη ερώτηση. Όπως ε, συμβαίνει συχνά, ε, πρόκειται για ένα δίλημα. Για την τελευταία σας ερώτηση. Μέχρι στιγμή ε, εγώ ξέρω μόνο μία έρευνα που είχε δημοσιεύσει ένας ε, γερμανός δικηγόρος για το Συμβούλιο της Ευρώπης που ασχολήθηκε με τον ορισμό του τι οικογένεια τι θα πει η ιδεολογική συγγένεια και όλοι αυτοί οι γενικοί ορισμοί και πράγματι έχουμε ένα δίλημα εδώ γιατί αφενός είναι γενικόλογοι και ευρύτατοι αυτοί οι ορισμοί και βεβαίως αλλάζουν η έννοια της οικογένειας αλλάζει η έννοια της υπηκότητας αλλάζει οπότε υπό μια έννοια θα πρέπει να έχουμε έναν πιο ακριβή ορισμό. Τι εννοούμε συγγενείς, ποιος ε, εμπίπτει στον ορισμό, τι εννοούμε οικογένεια. Αλλιώ θα είναι ευρύτατοι οι ορισμοί. Από την άλλη, ε, δηλαδή, τι που θέλουμε να πάμε, ε, σε, ως ποιο βαθμό. Αν θέλουμε με την οικογένεια να καλύψουμε το θείο μου στην Αμερική. Ε, δηλαδή μπορεί να πάει πολύ μακριά ο ορισμός της οικογένειας και τελικά θα καταλήξουμε σε παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, σε απίστευτη γραφειοκρατικοποίηση της πολιτικής ε, σύγκρουσης συμφερόντων. Είναι δίλημα λοιπόν αφενός χρειάζεται ένας καλύτερος ορισμός Αλλιώς το άρθρο 57 είναι άχρηστο. Από την άλλη, αν έχουμε πολύ λεπτομερείς ορισμούς, τότε θα μπούμε σε ζητήματα ιδιωτικής ζωής ε, και επίσης άρα μπορεί να είναι άχρηστα, ορισμοί αν καλύψουμε το θείο στην Αμερική όπως σας είπα από μεταβία στο ξέρω. Προτείνω λοιπόν να μπει ένας αστερίσκος ε, στο κείμενο ε, για το τι εννοούμε. Να έχουμε έναν ακριβή ορισμό της οικογένειας, αλλά πάντα έχοντας κατά νου ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε πολύ μακριά και σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειες, αλλιώς ε, θα βλάψουμε άλλα πράγματα τα οποία θεωρούμε σημαντικά. Κώδικες ε, συμπεριφοράς και δεοντολογίας. Ας επανέλθουμε στο ζήτημα της εμπιστοσύνης. Δύσκολο μπορούμε να προτείνουμε βέλτιστες πρακτικές. Βρήκαμε ενδιαφέρουσε βέλτιστες πρακτικές, ε, είπαμε την Ορβηγία, η Ολλανδία επίσης. Όλα αυτά υπάρχουν στην έρευνα. Αλλά το να προτείνουμε κάτι τέτοιο είναι πάντα δύσκολο. δύσκολο. Και σχετίζεται ακριβώς με το ζήτημα αυτό της εμπιστοσύνης. Σε γενικές γραμμές αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι χώρες εκείνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το υψηλότερο επίπεδο διαφοράς έχουν και υψηλό επίπεδο δυσπιστίας στο πολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς θεσμούς και ταυτόχρονα έχουν τους πιο λεπτομερείς κανόνες που υπάρχουν. Επίχει η Βουλγαρία έχουν ένα φανταστικό τέτοιο σύστημα, το οποίο είναι φανταστικό στη θεωρία. Ταυτόχρονα οι χώρες αυτές έχουν υψηλά επίπεδα διαφθοράς. Από την άλλη αναφέρατε τις χώρες της ε, Σκανδιναβίας χώρες με χαμηλά επίπεδα διαφθοράς. Δεν μιλάω για σύγκρουση συμφέρονο γιατί είπατε δεν το ξέρουμε αυτό. Υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και χαμηλό επίπεδο ρύθμισης. Και αυτό όταν πάει κανείς στην ε, Σκανδιναβία Ίσως αυτό δεν απαιτείται γιατί υπάρχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνη. Ανέφερα ότι οι πολιτικές αυτές ε, συγκρούσεις συμφερόντων είναι πολιτική δυσπιστίας. Οπότε δεν ξέρω εάν μπορεί τώρα να επαναληφθεί το μοντέλο αυτό με υψηλ... σε χώρες με υψηλά επίπεδα δυσπιστίας. Αυτό μας δείχνει ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων πάντα πρέπει να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες. Και για να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπα στην αρχή, εγώ είμαι πολύ προσεκτικός για να προτείνω βέλτιστες πρακτικές. Γιατί οι λόγοι για διαφθορά, για σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να είναι πολύ και διαφορετική και σχετίζεται με την κάθε κουλτούρα, την διοικητική κουλτούρα της κάθε χώρας για το θέμα του κώδικα. Εδώ θα είμαι σύντομος. Ε, οι ειδικοί στον τομέα της διαφθοράς ε, πάντα ξεκινάνε με μια διαφοροποίηση. Το μιλάνε για μη δεοντολογική συμπεριφορά. Λένε πως οι λόγοι μπορεί να είναι ατομικοί, προσωπικοί του καθενός. Αν θέλει κάποιος να είναι κακός, είναι κακός. Αν θέλει να κάνει κάτι αντιδιοντολογικό θα το κάνει. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι που οφείλονται στην κουλτούρα ενός οργανισμού ε, και κοινωνική ρόλη ε, πολιτισμική κτλ. Χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνη. Έχει αποδειχτεί ότι αήπια μέσα όπως οι κώδικες ε, δεοντολογίας χρησιμεύουν. Εγώ είμαι υπέρ των κωδίκων δεοντολογίας αλλά δεν είναι αποτελεσματική για τα άτομα εκείνα τα οποία σκεμμένα θέλουν να συμπεριφερθούν αντιδιοντολογικά. Μπορεί να χρησιμεύουν για τα άτομα εκείνα τα οποία θεωρούν τέτοιου κώδικες ως χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές ε, που προωθούν μια κουλτούρα κτλ. Αλλά για τα άτομα εκείνα τα οποία σκεμμένα παραβιάζουν τις ε, νόρμες αυτές είναι αναποτελεσματικοί οι κώδικες ε, διοντολογίας. Ίσως επίσης άρχισα κάπως ε, υπερβολική κριτική όταν μιλάμε για την αποτελεσματικότητα νομικά δεσμευτικών κανόνων. Όχι. θεωρώ ότι η αποτελεσματικότητα πρέπει να πηγαίνει κατά περίπτωση ανά χώρα, ανά κλάδο Γι' αυτό είναι περίπλοκο το ζήτημα και ποτέ δεν θα έλεγα ότι οι νόμοι κυρώσεις ε, μια συμπεριφορά που βασίζεται στη συμμόρφωση είναι αναποτελεσματική. Όχι, χρειάζεται, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε ήπια μέσα και χρειαζόμαστε ήπια μέσα και βεβαίως και νομοθεσία, αλλά και ένα τελείως καινούργιο μενού ψυχολογικών μέσων. Π.χ. μιλήσαμε για τη χαμηλού επίπεδου όχληση. Ε, ε, επίσης η ψυχολογία παίζει ένα σημαντικό ρόλο Γερμανοί π.χ. δεν θέλουν να συζητούν αυτό το ζήτημα, όχι γιατί α, το, δεν τους απασχολεί, αλλά θεωρούν κάτι, θεωρούν κάτι το οποίο εντάξει δεν είναι σοβαρό, δεν, δεν τους απασχολεί, είναι κάτι το περίεργο. Ε, αυτό δεν λύνεται με νόμους. Ε, χρειαζόμαστε νέα μέσα. Το θα ασχοληθώ πολύ σύντομα με το πρόβλημα που θέσατε στη δεύτερη ερώτησή σας για τις αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά και είναι το δύσκολο στο πολυπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακριβώς γι' αυτό μιλάμε. Έχουμε να κάνουμε με κοινή διαχείριση όπου η εφαρμογή είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και όπως έδειξε η μελέτη πιστεύω πως η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των κρατών μελών τώρα η σύγκρουση συμφερόντων και η αντίστοιχη πολιτική, το πλαίσιο που θεσπίστηκε από το ευρωπαϊκό επίπεδο, το επίπεδο της Ένωσης, είναι κατάλληλο και παρκές. Τα προβλήματα σχετίζονται με τις διαφορές και τη μεγάλη ποικιλία και τις μεγάλες διαφορές της εφαρμογής. Αυτό είναι που δυσχεραίνει το όλο ζήτημα. Σε ένα ενιαίο κράτος δεν θα υπήρχε μια τέτοια κατάσταση. Τώρα, όπως ακούσαμε, εν ναι, είχαμε διαφορετικές προσεγγίσεις στο ατομικό επίπεδο, στο επίπεδο διακυβέρνησης, υπάρχει δημιουργία ικανοτήτων, υπάρχει εκμάθηση, δημιουργία κατανόησης και υποδομής για την αντιμετώπιση ζητημάτων. Αλλά επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένας κυρωτικός μηχανισμός. Και πιστεύω πως συμφωνούμε στο γεγονός πως οι χώρες αποδέκτες οφείλουν να λογοδοτήσουν στην κοινότητα από την οποία λαμβάνουν. Γι' αυτό και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα δικαίου, χρειαζόμαστε μια κοινή κατανόηση των νομικών κυρώσεων ως τελευταία λύση, αν θέλετε. Ένα συνδυασμό είναι και πάλι καλό. Χρειαζόμαστε ελάχιστα νομικά πρότυπα τα οποία θα πρέπει να επιβάλλονται και θα πρέπει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μια κουλτούρα βιωσιμότητα ε, που αποτελεί και μέρος απάντησης στην πολύ δύσκολη ερώτηση νούμερο ένα. Πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στη διοίκηση και στο πολιτικό σύστημα. Πιστεύω πως αυτό σχετίζεται με το γεγονός πως οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν πως εκείνοι που έχουν την εξουσία οφείλουν να λογοδοτούν σε αυτούς. Όσο υπάρχει παρέτηση, δηλαδή όσο ο κόσμος πιστεύει πως αυτοί εκεί πέρα κάνουν έτσι ούτως ή άλλως ό,τι θέλουν, τότε δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να γίνει σε συστημικό επίπεδο. Πρέπει να επιτευχθεί ένας διάλογος, μια διαδικασία διαλόγου και νομίζω πως ήθελες να προσθέσεις κάποια πράγματα ακόμα. Είπε πολύ σημαντικά πράγματα ο συνάδελφος, αλλά από πλευράς Πολωνίας να σας πω πώς τα βλέπουμε, γιατί είχα αναλάβει τα σχετικά στη χώρα μου και θα πρέπει να συμφωνήσω 100% με είπε ο Κρίστοφ, ότι η σύγκρουση των συμφερόντων βασικά έχει να κάνει με καθημερινά ζητήματα. Δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Οπότε και όσον αφορά τη διοίκηση, τελικά είναι το να μην ευαισθητοποιείται κανείς το φαινόμενο και συνέπειες του. Υπάρχουν ένα σωρό νόμοι σχετικά σε επίπεδο εθνικού δικαίου για την σύγκρουση των συμφέροντων στα πλαίσια της δημοσιοπαραγγελίας, στα πλαίσια της διοίκησης. Ένα σωρό εθνικοί νόμοι υπάρχουν. Υπάρχει βέβαια και η αυτορύθμιση. Κάτι που καθιερώθηκε από κάποιες ε, αρχές, κάποιες κώθηκες στην δηλαδή. και άλλοι σε ιστορικής λειτουργίες. Όμως αποδείχθηκε από τη μελέτη του 14 νομίζω ότι ακόμη δεν υπάρχει επίγνωση του φαινομένου. Τι πάει να πει σύγκρουση συμφερόντων, σε τι συνίσταται και τι πρέπει να γίνει για να προλάβουμε το κακό. σχετικοί κανόνες αφορούν πολλές κατηγορίες ε, υπαλλήλων. Συνήθως αφορούν ε, δημοσίους υπαλλήλου, αλλά υπάρχουν και άλλοι κανόνες ε, για την αυτοδιοίκηση, ας πούμε. Βέβαια και θέμα εκπαίδευση, κατάρτιση, ιδίω για εκείνου που ασχολούνται με τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, χωρίς να είναι υπάλληλοι. Ε, εργολάβοι, συμβασιούχοι. Πολύ σημαντικό. Γιατί το περασμένο μήνα ενέκρινε το Κοινοβούλιο το κείμενο για την προστασία των πληροφοριδιωτών, καταδοτών, και αυτοί πρέπει να καλυφθούν. Εμπειρογνώμονες, δικαιούχοι, διάφοροι που βρίσκονται εκτός δημόσιας διοίκησης. Γιατί τα προβλήματα της σύγκρουσης συμφερόντων τους αγγίζουν. Θα πρέπει να το δούμε ευρύτερα το θέμα. Ξέρω ότι η μελέτη επικεντρώθηκε στις ε, εποπτικές ελεγκτικές επιτροπές. Αλλά θα πρέπει να δούμε γενικότερα τι ισχύει με την ε, πολιτική κατάσταση διαφθοράς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντική και για το θέμα μας. Ευχαριστώ πολύ ο συνάδελφος Μπόγκιν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ερώτηση ή σχόλιο, θα το δώσω στο τέλος της παρέμβασής μου. Θα αρχίσω βλέποντας ότι είναι σημαντικό να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς στο σχεδιασμό και στην παροχή διαθροτικών ταμείων, είτε είναι ο δημόσιος, ο ιδιωτικός τομέας, η ΜΚΙΟ ή άλλοι τομείς, σημαντικό για τα διαφορετικά ταμεία είναι η εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων ταμείων, τομέων, συγγνώμη. Και πιστεύω πως πρέπει να το ενθαρρύνουμε. Η εμπειρία δείχνει πως δεν υπάρχει έλλειψη κωδίκων κανόνων και οι περισσότεροι άνθρωποι που συμμετέχουν στις επιτροπές αυτές γνωρίζουν τους κανόνες αυτούς επειδή όταν γίνεται κανείς μέλος μιας επιτροπής ή ενός συμβουλίου γίνονται μαθήματα εισαγωγής όπου εξηγούνται οι κανόνες σε σχέση με τις συγκρούσεις Το Μεγαλύτερο ερώτημα είναι η παρακολούθηση των κωδίκων δεοδολογίας όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερώτημα. Ακούγοντας τον Κρίστοφ και τον Τόμας, από ό,τι φαίνεται λέτε δύο πράγματα, τα οποία είναι διαμετρικά αντίθετα. Νομίζω ο Κρίστοφ έθεσε το βάρος στον πρόεδρο των διάφορων επιτροπών συμβουλίων και αυτό πιστεύω πως θα είναι αρκετά δύσκολο στην πραγματικότητα, επειδή το είπε και εσύ ο ίδιος. Οι πρόεδροι αυτοί είναι άνθρωποι με διαφορετικά επίπεδα εμπειρία, διαφορετικές προσωπικότητες. Κάποιοι ίσως είναι... έχουν περισσότερη τάση να ασχοληθούν με το ζήτημα των ε, συγκρούσεων συμφερόντων και ο Τόμας πέρασε στο άλλο άκρο μιλώντας για περισσότερη παρακολούθηση, περισσότερη λεπτομερή καταγραφή, αλλά θα χρειαστούν περισσότεροι υπάλληλοι επίσης. Και μπορώ να το πω από την οπτική γωνία τη περιφερειακή ανάπτυξη. Και αυτό είναι το τελευταίο που χρειάζονται τα διαρθρωτικά ταμεία. Αν μιλήσει κανεί με οποιονδήποτε από τον τομέα αυτό, των διαφορετικών των ταμπίων, όλοι θα σας πούν, ζητούν περισσότερη απλούστευση και όχι περισσότερη παρακολούθηση. Πιστεύω πως πρέπει να φέρουμε τα δύο άκρα αυτά σε μια ισορροπία. Στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού πρέπει να βρούμε έγκαιρα έναν μια ισορροπία. Κατά πόσον τα χρήματα ξοδεύονται με τον σωστό τρόπο, με τήρηση όλων των κανόνων, συμπεριλαμβανομένων αυτών περί σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά επίση δεν πρέπει να μπει υπερβολικό αριθμό κανόνων έτσι ώστε οι ωφελούμενοι, οι ενδιαφερόμενοι να αποθαρρυνθούν από τη συμμετοχή. Πρέπει να βρούμε την χρυσή τομή. Πιστεύω πως πρέπει να έχουμε τους ε, κανόνες αντιμετώπισης κινδύνων, οι οποίοι ισχύουν επίσης για τη σύγκρουση συμφερόντων. έχουμε εφαρμογή των κανόνων για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Αν υπάρχουν οργανισμοί ή αρχές που είχαν προβλήματα στο παρελθόν ή που έχουν εκφράζουν την ανησυχία τους, τότε πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας σε αυτούς. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία σωστά. Πιστεύω πως η απάντηση είναι ότι πρέπει να κινηθούμε κάπως στο ενδιάμεσο έβαλα και τον εαυτό μου στον κατάλογο των ομιλητών. Θα ήθελα να μιλήσω για μια περίπτωση από ένα κράτος μέλος όπου ένας δημοτικός σύμβουλος, αμυστή δημοτικός σύμβουλος, ήταν μέλος ενός ε, συμβουλίου το οποίο ανοίγει τις προσφορές από τον κλειστό φάκελο. Και ως μέλος της ομάδας αυτή ανακάλυψε πως η δική του εταιρεία είχε υποβάλει προσφορά και η δική του εταιρεία στην οποία εργαζόταν Εκεί διαφέρουν οι διάφορες εκδοχές. Οι μεν λένε ότι κατευθείαν αποσύρθηκε, εγκατέλειψε το χώρο. Στο τέλος έγινε μια εξέταση, διερεύνηση για σύγκρουση συμφερόντων και ο άνθρωπο αυτός στο τέλος δεν έχασε μόνο τη θέση εργασία του, αλλά αναγκάστηκε να μετακομίσει σε μια άλλη πόλη. Επειδή η δημόσια αντίδραση στο φαινόμενο αυτό ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να συνεχίσει να ζει στην πόλη αυτή. Απευθύνθηκε σε μένα, μου το ανέφερε, γνωρίζω μόνο τη μία εκδοχή, τη δική του. Πιστεύω πως χρειαζόμαστε κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες για την πράξη. Η μελέτη σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να γράψουμε μέσα στους κανονισμούς για τα διαφορετικά ταμεία που θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και όχι υπερενέργειες. Αν μπορούσατε να ασχοληθείτε λίγο με αυτό, δεν είναι ζήτημα αριθμού κανόνων, αλλά της σαφήνειας και της εφαρμογής τους. Εκεί συμφωνούμε. Βλέπουμε πως μερικά κράτη-μέλη έχουν κατακαιρματισμένη νομοθεσία όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων. Είναι η περίπτωση που ανέφερε η Μαρτίνα όταν υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Έχουμε κυβερνήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου μέλη των κυβερνήσεων έχουν μερικές απασχολήσεις. Ε, αυτή είναι μια κατάσταση η οποία προκαλεί για φαινόμενα παντός είδους. Σκέφτομαι ένα κράτος μέλος στη Νότια Ευρώπη, εκεί υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Το ισπανικό παράδειγμα έχει ενδιαφέρον Όσον αφορά τις παρατυπίες με την Ισπανία έχουμε μεγάλα προβλήματα. Δεν θέλω να τα συσχετίσω τα δύο, αλλά προκαλεί την προσοχή. Τι μας συστήνεται, έχετε τον λόγο. Ο συνάδελφος Τσέλερ, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε από την δική μου την εμπειρία στην Γερμανία. Αυτά τα ρυθμίζει νομίζω κώδικας, ο οποίος, ε, ο νόμος ο οποίος καθορίζει τα της διοίκησης. Ε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο ε, μπορεί να κάνει κάποιος εντάξει και εμένα ή όχι Μα έχει το τι προβλέπει ο νόμος και βεβαίω εδώ πέρα αν κάνουμε μια σύγκριση των νομοθεσιών των σχετικών στι 28 χώρες να δούμε πώς θα ρυθμιστεί. Λοιπόν, δεν, δεν υπάρχει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παλεύουμε εμεί. Η Κομισιόν αμήνεται βεβαίω ε, με νύχια και με δόντια. Κύριο Τάκουλα, σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει κάποια ελάχιστη ευρωπαϊκή ρύθμιση ή τουλάχιστον μια πρόταση γιατί υπάρχουν ε, διαφορές στα κράτη-μέλη. Καταπολεμούμε βεβαίω ε, και την ε, διαφθορά και αυτό απαιτεί, όπως είπαμε, κάποιες συζητήσεις για το ποια είναι η γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μπορούν οι εταιρείες συγγενών ε, να λάβουν μέρος σε ένα διαγωνισμό, σύζυγοι, ξαδέρφια, ποιος επιτρέπεται και ποιος όχι. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρους ε, κανόνες, γιατί γνωρίζουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη ε, μπορούν να κάνουν οι συγγενείς ό,τι θέλουν. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Μα το θέμα δεν είναι μόνο γιατί αναφέρθηκαν παραδείγματος χάρη και κάποιες ε, επιτροπές ε, κατευθυντήριες ε, ή αυτές οι οποίες εφαρμόζουν τα διαρθρωτικά ταμεία. Τι κάνω εγώ εάν είναι να δώσω να αναθέσω έναν διαγωνισμό και είναι τόσο χαμηλά τα κατόφλια ώστε ε, φτάνω αμέσως ε, στο ότι πρέπει να είναι πανευρωπαϊκή η προκήρυξη του διαγωνισμού. Κάτι το οποίο είναι πρόβλημα για πολλούς Δήμους βεβαίως. Ταυτόχρονα η περιφέρειά μου ή το κρατήδιο λέει ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την περιφερειακή μας η οικονομία και θα πρέπει να προτιμηθούν ε, τοπικές εταιρείες. Εκεί πέρα έχω μπλέξει, βρίσκομαι αφενός μεταξύ των ευρωπαϊκών κανόνων και των πολιτικών απαιτήσεων της ε, περιφέρειας. Που τελικά μια που οι ΟΤΑ συνήθως βεβαίως διοικούνται από αιρετούς ε, θέλουν να ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Ε, αυτή είναι μια κλασική περίπτωση σύγκρουσης και πρέπει ακριβώς ε, να προσπαθήσουμε, προσπαθεί κανείς να βρει μια ισορροπία κατά τη, και μια αιτιολόγηση κατά τη σύνταξη της προκήρυξης. Θα ήθελα να δώσω και τον λόγο στην ε, Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιου, στην κυρία Ντελαφράγκα. Παρακαλώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να σας πούμε δύο λόγια και από πλευράς μας. Πρώτα-πρώτα ε, θεωρούμε από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής αυτή την μελέτη, τη θεωρούμε πολύ ενδιαφέρουσα και οπότε ε, χρειαζόμαστε λίγο χρόνο τόσο ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο, να εξετάσουμε όλες τις συστάσεις, να δούμε ακριβώς τι συμπεράσματα βγαίνουν, τι συνέπειες μπορεί να υπάρξουν, τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τις ε, πρακτικές επί τη βάση των συστασιών σας. Επίσης να σας αναφέρω ότι δεν θέλω να ακολουθήσω ε, αμυντική γραμμή πλεύσης. Ε, δεν θεωρώ ότι αυτή η μελέτη αποτελεί μια επίκριση ε, για το τι ισχύει, για τους κώδικες, για τους κανόνες, για τους νομοθεσίες. Το αντίθετο, το αντίθετο. Λέμε ότι υπάρχουν αρκετοί κανόνες, αρκετή νομοθεσία, αρκετοί κώδικες. Οπότε το θέμα είναι το ότι έχουμε ένα περίπλοκο ζήτημα, μια δύσκολη έννοια όπως την σύγκρουση συμφερόντων και το θέμα είναι ακριβώς πώς θα εποπτεύσουμε, πώς θα ελέγξουμε το τι γίνεται. Ε, αυτό γίνεται στα κράτη-μέλη και εμείς θέλουμε να δούμε τι γίνεται σε κάθε χώρο, στην πραγματικότητα, πώς μπορούμε να έχουμε τις ε, άριστες των πρακτικών για να χειριστούμε την κατάσταση. Τα ξέρουν οι ασχοληθέντες με την μελέτη και οι ευρωβουλευτές τι ισχύει. Δεν τα επαναλάβω. Ε, τι γίνεται με την ε, πρόληψη, ανείχνευση και διόρθωση σε σχέση με τα ταμεία. Αλλά να σας πω κάτι άλλο. Ιδίω όσον αφορά την σύγκρουση συμφερόντων στις εποπτικές ε, επιτροπές. Αυτό είναι κάτι το νέο. Τα έχουμε συζητήσει. Μέτρα κατά της απάτης. Μέτρα κατά της σύγκρουσης συμφερόντων. Τι γίνεται με τις δημόσιες συμβάσεις για τα επενδυτικά ταμεία. Ε, τι γίνεται με την ε, διοίκηση, με αυτούς που από πλευράς δημόσιας διοίκησης διαχειρίζονται τα ταμεία και τους πόρους. Εγώ έχω διαλέξει κάποια κρατημέλη με τα οποία συνεργάζομαι για τα ταμεία και τους πόρους αυτούς και προσπαθώ να πετύχω μια εύρεθμη λειτουργία των επιτροπών. Θέλω τα προγράμματα να σχεδιάζονται και να εποπτεύονται όχι μόνο από την κεντρική διοίκηση, αλλά από όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους, τις μη κυβερνικές οργανώσεις. Ε, δύσκολο ήταν, ε, ιδίω σε κάποιες περιπτώσεις, να εξασφαλίσουμε το ότι αυτές οι υποπτικές επιτροπές αποτελούν ένα βήμα που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και που όλα συζητούνται όπως πρέπει. Επίσης βέβαια υπάρχει η ενδυνάμιση σύγκρουση συμφερόντων όσο περισσότεροι εμπλεκόμενοι συμμετέχουν σε μια επιτροπή ε, τόσο πιο πιθανό είναι να συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων οπότε ιδίω εμείς ως περιφερική πολιτική θα πρέπει να προσέξουμε τα εξής παγκόσμιες άριστες πρακτικές. Ε, δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε να δανειστούμε κάτι που αποδίδει σε μια περιφέρεια, να το μεταμοσχεύσουμε αλλού. Αυτό είναι η ομορφιά, αυτό είναι και όμως και η δυσκολία της δουλειάς μας. Όποτε αναδύεται ένα πρόβλημα, θα πρέπει κανείς να ε, σκεφτεί τι μπορεί να ισχύσει, που είναι το καλύτερο για τη συγκεκριμένη περιοχή, περιφέρεια και έχουν πολλές φορές κάποια άλλα ε, μέσα πολιτικής, τα λεγόμενα peer to peer, όπου εμπλέκονται ισότιμοι και αυτό σχετίζεται και με την πρόληψη στις επιτροπές, πρόληψη του φαινομένου. δεν είναι κάτι που άπαξ επισημαίνεται και μαθαίνεται η σύγκρουση συμφερόντων. Θα πρέπει κανείς να περνά από κύκλους α, εκπαίδευσης και εκμάθησης. Αυτό και κάνουμε. Αυτή η κύκλη εκπαίδευσης, εκμάθευσης, συνειδητοποίησης. Επίσης, Πρόσφατα έγινε μια μελέτη που την αναφέρατε και εσεί για την πρόληψη της απάτης και τη διαφθορά στα επενδυτικά ταμεία τη Ένωση. Εισετάστηκε και η πρόληψη της σύγκρουση των συμφερόντων. Το τονίσατε και εσείς, πολύ σημαντικό, το πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα κατά της απάτης πόσο αποτελεσματικά γίνεται η εποπτεία. Άρα δεν κοιτάμε τις διαδικασίες και τα, τις, τους κανόνες, αλλά το πόσο αποτελεσματική γίνεται η εποπτεία. Άρα κοιτάμε τα αποτελέσματα, τη λειτουργία τους των κανόνων κλπ. Και, όχι το αν υπάρχουν κανόνες. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ. Όλα αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε και θεωρείτε ότι χρειάζεται, Πρόεδρε, να τα ξανασυζητήσουμε για το τι πρακτικά συμπεράσματα θα εξαγάγουμε από όλα αυτά. Ευχαριστώ και ο πάρα πολύ. Πιστεύω πως θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επί του θέματος. Δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος. Θα συνεχίσουμε στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ. Να, να ρωτήσω, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.